Ε, τώρα είναι οι ερωτήσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίασή σας κύριε υποψήφια αντιπρόεδρε. Και τώρα θα περάσουμε στον πρώτο γύρο παρατηρήσεων και ερωτήσεων. Εκ μέρους των πολιτικών ομάδων καταρχήν, ο κύριος Κάριμς εκ μέρους του ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σεύκοβιτς. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε τι θα πρέπει να σημαίνει να εξηγηθεί κανείς εντός πέντε ημερών με ένα εντελώς νέο χαρτοφυλόκιο. Νομίζω ότι όλοι εδώ κατανοούμε την κατάσταση στην οποία βρεθήκατε. Ωστόσο θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι σε σχέση με την ασφάλεια του εφοδιασμού. Όπως ξέρετε και όπως είπατε, εμείς εξαρτώμαθα πάρα πολύ στις εισαγωγές ενέργειας πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ τη μέρα. Και ο τομέας του αερίου θέτει πάρα πολλές προκλήσεις γιατί είναι δύσκολη η μεταφορά μέσω αγωγών. Επίσης, στον τομέα του αερίου έχουμε μια όλο και μεγαλύτερη εξάρτηση από την παροχή από την αερίου από τη Ρωσία. Και εσείς ο ίδιος αναφέρατε ότι ε, η Ουκρανία, χρησιμοποιείται σαν ε, όπλο. Δύο ερωτήσει. Εσείς ως ε, Επίτροπος θα υποστηρίξετε τον αγωγό South Stream ο οποίος θα αυξήσει την ανεξαρτησία από την Ρωσία και δεύτερον πώς προτείνετε να μειωθεί η εξάρτησή μας από την Ρωσία και να αυξηθεί συνολικά η ασφάλεια εφοδιασμού. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τις δύο ερωτήσεις που είναι απολύτως ε, ε, σημαντικές και θα καθορίσουν το έργο μου τα προσεχή πέντε χρόνια. Θα Ερευνητά καταρχήν στο South ε, Stream, το οποίο, έχει, το οποίο η λειτουργία έχει ανασταλεί. Και επειδή δεν μπορούμε να αποδεχθούμε ένα τόσο μεγάλο έργο να γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω μιας εταιρεία η οποία δεν σέβεται τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Είναι λοιπόν απολύτως σαφές ότι εδώ θα πρέπει να έχουμε δύο βασικές ερωτήσεις που πρέπει να διευκρινιστούν. Πρώτον, μια απόλυτη προσήλωση προς τους ευρωπαϊκούς κανόνες και δεύτερον αυτό το οποίο περιγράφεται πολύ καλά στο, στη στρατηγική για την Ευρωπαϊκή Ενέργεια και Ασφάλεια πώς αυτό θα βοηθήσει την αύξηση επίπεδα ασφάλεια στην Ευρώπη, πώς δηλαδή θα διαφοροποιηθούν οι πηγές μας ενέργειες. Και για να είμαι ειλικρινής, δεν βλέπω το εγχείρημα αυτό πραγματικά να πληρεί αυτά τα κριτήρια. Γι' αυτό πιστεύω ότι μελλοντικά θα στρέψουμε ε, τις προσπάθειές μας και τις επενδύσεις μας προς τον νότιο διάδρομο. Νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό γιατί θα μας βοηθήσει να διαφοροποιήσουμε τις πηγές ενέργειας, να να πάρουμε αέριο από την Κασπία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και να έχουμε τη δυνατότητα να μην περιοριζόμαστε στις πηγές ε, του Αζερβαϊτζάν ε, φυσικού αερίου, αλλά ενδεχομένω να αναπτύξουμε μια καλή συνεργασία, ούτως ώστε να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις και με άλλη σημαντική πηγή, ε, το Τουρκμανιστάν. Η ξεκάθαρη προτίμησή μου λοιπόν να υπάρξει μια διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να έχουμε τα έργα για τον νότιο διάδρομο να εξελιχθούν και να τα υποστηρίξουμε πολιτικά πλήρως. Ευχαριστούμε πολύ εκ μέρους των σοσιαλιστών η κυρία Καθλίν Βαν Μπέμπτ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πίτροπε. Έχω κρυώσει και η φωνή μου είναι λίγο βραχνή. Ε, θα ήθελα να σα ρωτήσω κάτι για την Ενεργειακή Ένωση στο σύνολό τη. Όπω ξέρετε, υπάρχουν ήδη διάφορε ερμηνείε και ε, ε, σε σχέση με την ε, προσπάθεια να γίνουμε ανεξάρτητα από τη Ρωσία. Αλλά ωστόσο αυτό δεν είναι αρκετό για τη δική μας ομάδα. Εσείς αναφέρετε πέντε συγκεκριμένους πυλώνες που νομίζω καλύπτουν ε, την πλειονότητα αυτού που ονομάζουμε Ενεργειακή Ένωση. Θα ήθελα να εστιάσω σε δύο βασικέ ερωτήσει. Εάν δούμε αυτού του πέντε πυλώνε, ποιε είναι, ποιες είναι οι δικέ σα βασικέ προτεραιότητε και ποια θα είναι τα συγκεκριμένα μέτρα που θα παίρνετε εσεί για τα προσεχή έτη. Ευχαριστώ πολύ για αυτές τις ερωτήσεις. Πιστεύω ότι βεβαίω για ορισμένε από αυτές τις προτεραιότητες μπορούμε να προγραμματίσουμε και να συνεργαστούμε και ε, νομίζω ότι ορισμένε από αυτές θα πάρουν σάρκα και οστά. Ε, θα δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων αύριο που θα έχει ο Αντιπρόεδρος κ και οι Ρώσοι και η Ουκρανοί εταίροι. Ελπίζουμε να βρεθεί μια συμφωνία και να αποφύγουμε μια δραματική κατάσταση όσον αφορά την παροχή αερίου το χειμώνα στην Ουκρανία και στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Ε, ανησυχώ βεβαίως ε, ε, για το θέμα αυτό και αυτή είναι η άμεση μας προτεραιότητα. Αλλά εάν βάλουμε αυτό παράμερα, εάν δούμε τι γίνεται από στρατηγική άποψη, νομίζω ότι η καλύτερη δυνατή προσέγγιση θα ήταν να προωθήσουμε όλους τους πυλώνες από κοινού γιατί υπάρχουν πολλά κοινά στοιχεία ε, ταυτόχρονα και ελπίζω ότι θα έχουμε γρήγορα φιλόδοξες αποφάσεις του Συμβουλίου. Αύριο θα εκπροσωπήσω την ε, Επιτροπή στο Συμβούλιο και πραγματικά αναμένω πραγματικά ε, θετικά αποτελέσματα και την προετοιμασία των Ευρωπαίων, τη συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών. Θα πρέπει να δούμε πώς ε, θα μεταφέρουμε αυτό το πακέτο στο νομικό πλαίσιο, στο νομοθετικό πλαίσιο. Και την άνοιξη θα προετοιμάσουμε τη δική μας ε, θέση για ε, το Παρίσι. Και βεβαίως... Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Είναι πολύ σημαντικό να επιλέξουμε τα προγράμματα όσον αφορά το εργαλείο για τη διασύνδεση της Ευρώπης και να υπάρξει μια σωστή διαδικασία επιλογής και διαγωνισμών, ε, προκήρυξης διαγωνισμών για το καλύτερο πρόγραμμα. Ε, θα πρέπει επίσης να εστιάσουμε την προσοχή μας σε θέματα της εσωτερικής αγοράς γιατί ξέρετε ότι ήδη έχουμε συμφωνήσει ότι το 2014 θα έχει ολοκληρωθεί η ενεργειακή αγορά στην Ευρώπη και γνωρίζετε το αποτέλεσμα. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί στο τέλος αυτού του χρόνου. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε ταχαίως. Ευχαριστώ. Η κυρία Τζούλη Γκέρλινγκ έχει το λόγο από του συντηρητικού και μεταρρυθμιστές. Καλώ ήρθατε κύριε Σεύκοβιτ. Μέσα στη δομή που έχει δημιουργήσει ο κύριος Γιούνκερ, ο αντιπρόεδρο για την ενέργεια παίζει ένα κομβικό ρόλο για να μπορέσει να επιβλέπει το έργο των επιτρόπων στα συγκεκριμένα χαρτοφυλάκια. Αλλά μέχρι στιγμή οι αντιπρόεδροι δεν έχουν δώσει συγκεκριμένα δείγματα γραφή σε σχέση με τον ε, ρόλο του. Έχουμε μια σημαντική αλλαγή Τώρα, σε σχέση με την ε, παρακολούθηση των θεμάτων που έχουν να κάνουν με την κλιματική αλλαγή. Έχουμε από τη μια μεριά τα θέματα στρατηγικής για την κλιματική αλλαγή που περιλαμβάνουν τα αέρια θερμοκήπιων, ενώ τα, οι άλλες εκπομπές δεν λαμβάνουν υπόψη σε αυτό το πακέτο. Δεν υπάρχει συνέργεια, δεν συμπληρώνονται μεταξύ τους αυτά τα δύο εγχειρήματα και οι ημερομηνίε δεν ταιριάζουν. Τα κράτη-μέλη λοιπόν δεν έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν εκτικού στόχου. Δεν είναι αυτή η καλύτερη νομοθεσία λοιπόν και πώ μπορείτε να το αντιμετωπίσετε το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γκέρλινγκ. Παρουσιάσετε μια κατάσταση που δεν ήταν και η βελτιότερη και γι' αυτό ο νέος πρόεδρος της Κομισιόν θέλησε να αλλάξει η δομή της Κομισιόν γιατί αυτό θα δημιουργήσει δυνατότητα συνεργασίας από την αρχή όλων των εγχειρημάτων, όχι μόνο για τους επιτρόπους αλλά και για τις υπηρεσίες τους. Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ο αρμόδιος ε, αντιπρόεδρος και οι αρμόδιοι επίτροποι να μπορέσουν να δώσουν το σωστό παράδειγμα συνεργασίας μεταξύ τους. Αν δείτε το νέο οργανόγραμμα της Κομισιόν, αυτή είναι η θέση που θα έχω αν με εγκρίνετε μετά από αυτή την ακρόαση και αυτοί είναι οι επίτροποι τους οποίους πρέπει να συνδενήσω. Σας τονίζω εδώ πέρα ότι το χρώμα που με αντιπροσωπεύει εδώ είναι πράσινο. Θα είναι πολύ σημαντικό να συνεργαστώ στενά με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες για τα θέματα της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Μπορώ λοιπόν να σας υποσχεθώ ότι από τη δική μου οπτική γωνία ο ρόλος του Αντιπροέδρου είναι ρόλος συντονιστή είναι αυτός ο οποίος πρέπει να εξασφαλίσει ότι συνεργάζονται όλες οι υπηρεσίες από την αρχή και έτσι δεν θα έχουμε μια υπηρεσία να ζητάει ένα σύνολο στόχων ενώ μια άλλη υπηρεσία έχει διαφορετικούς στόχους ή έχουν διαφορετικά συστήματα για να παρέχουν αναφορές η κάθε υπηρεσία. Και έτσι όταν φτάνουμε στο καταληκτικό στάδιο, στο σώμα των επιτρόπων, δεν θα υπάρχουν προβλήματα συγκρούσεων γιατί το, το γραφείο κάθε επιτρόπου προσπαθεί να φέρει τα πράγματα προς τη μια προς την άλλη μεριά. Είναι δύσκολο λοιπόν στο τελικό στάδιο να αντιμετωπιστούν όλα αυτά. Θέλουμε να αναστρέψουμε αυτή τη λογική, θέλουμε από την αρχή να υπάρχει συνεργασία και συντονισμός ώστε να εξασφαλίσουμε ότι πράγματι προχωρούμε από κοινού και να εξασφαλίσουμε επίσης ότι δεν θα χρειάζεται να υπάρχει περιττή γραφειοκρατία και παράδοση εκθέσεων και υπερβολικές υποχρεώσεις για εκθέσεις όπως το παρελθόν. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος ε, Φέντερ λέει <clears throat> από την ε, φιλελεύθερη ομάδα είναι και αντιπρόεδρο μας. Σας ευχαριστώ κύριε πρόεδρε και κύριε υποψήφια επίτροπε. Εδώ είμαι. Έχω πάρει νέα γραφεία στο γραφείο μου ώστε όταν ξανάρθετε να με επισκεφτείτε θα είσαστε πιο άνετα. Εσείς ουσιαστικά έχετε απαντήσει στο πρώτο ερώτημά μου που είναι πώς θα μπορέσετε να γίνετε μια πρωτοπόρα να γίνει η Ευρώπη πρωτοπόρα δύναμη στι ανανεώσιμε ενέργειε. Υπάρχει συνεχή συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη γεωπολιτική, για την οικονομική ανάπτυξη και για την ανανεώσιμη ενέργεια. Ένα από τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα σημείο όπου θα πούμε ότι η οικονομική ανάπτυξη δεν θα πρέπει να αναχαιτίζεται από την ανάγκη αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Θα ήθελα να πείτε λίγο περισσότερα για το θέμα αυτό. Βλέπετε την ε, αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής να απειλεί την οικονομική ανάπτυξη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ πολύ για το ερώτημα. Δεν το πιστεύω ότι υπάρχει σύγκρουση. Πιστεύω ότι και η βιομηχανία η βιομηχανική ανάπτυξη και μια ανταγωνιστική πολιτική για την πράσινη οικονομία πρέπει να αλληλοϊποστηρίζονται. Εσείς είσαστε στις επιτροπές σας οι αρμόδιοι για τα θέματα περιβάλλοντος ενέργειας και ξέρετε πολύ καλά ποιο είναι το τίμημα των εισαγωγών ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε πόσο μεγάλη είναι η αστάθεια που αντιμετωπίσουμε. Και αυτό γίνεται ουσιαστικά κάθε φθινόπωρο. Αναδύεται πάλι αυτό το πρόβλημα γιατί εξαρτώμαστε πάρα πολύ από ενεργειακές πηγές έξω, της, έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι. Οι εναλλακτικές ενέργειες μας δίνουν λοιπόν εγχώρια ενέργεια. Είναι κάτι το οποίο η ηλιακή ενέργεια, η αιωλική ενέργεια κτλ. Όλα αυτά μπορούμε να τα έχουμε στην Ευρώπη και οι εταιρείε μας είναι οι πρωτοπόροι σε παγκόσμιο επίπεδο για τις τεχνολογίες αυτές ανανεώσιμων ενεργειών και είναι πάρα πολύ επιτυχημένες και σε άλλες αγορές, σε χώρες όπως είναι η Κίνα όπου αρχίσουν να καταλαβαίνουν και εκεί οι πολίτες ότι δεν έχει νόημα να τρέξει μαραθώνιο φορώντας μια μάσκα επειδή είναι μολυσμένη η ατμόσφαιρα και δεν έχει νόημα να κλείνεται βιομηχανίες για να μπορούν να βλέπουν οι θεατές στους Ολυμπιακούς Αγώνες ποιος τρέχει σε ποια διαδρομή. Είναι απαραίτητο λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι θα μπορούμε να έχουμε μια πρόοδο και θα δώσουμε ένα σωστό πλαίσιο και ένα καθεστώς νομικής ασφάλειας στις επιχειρήσεις, στη βιομηχανία, ώστε να προωθήσουμε τις πράσινες τεχνολογίες με έναν τρόπο ο οποίος δεν αποτελεί εμπόδιο για την ανάπτυξη της βιομηχανίας, αλλά δίνει προσιτή και καθαρή ενέργεια, πράσινη ενέργεια, η οποία θα βοηθήσει και την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Σιλικιώτης από την ΚΟΕ. Κύριε Αντιπρόεδρε, στην ανακοίνωση της Κομισιόν με θέμα την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ενεργειακή Ασφάλεια δεν υπάρχει καμία ουσιαστική αναφορά στα μεγάλα κοιτάσματα που έχουν ανακαλυφθεί στην Ανατολική Μεσόγειο και ο σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσουν για την ενίσχυση τη ενεργειακή ασφάλεια, ούτε στην εισαγωγική σα τοποθέτηση, κύριε Σεύκοβη, αναφερθήκατε σε αυτά ε, τα κοιτάσματα. Ε, αναφέρεστε μόνο γενικά στη δημιουργία ενός μουσιακού κόμβου. Ε, πώς αντιλαμβάνεστε τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσουν αυτά τα κοιτάσματα και ιδιαίτερα τα κοιτάσματα που ανεβρέθηκα στην Κύπρο να πω ότι τώρα ε, προχωρούν οι ευρωπαϊκές εταιρείες σε σημαντικές φιλόδοξες ερευνητικές γεωτρήσεις. Είναι στις προτεραιότητες σας ακριβώς να αναπτυχθεί ένας μεσογειακός κόμβος μέσω διαδρόμου από την νοτιοανατολική Μεσόγειο προς την Ευρώπη και θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί έναν έργο για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας σε αυτήν την περιοχή. Thank Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ένα πράγμα το οποίο αναφέρθηκε στις ε, πρώτες μου παρατηρήσεις αλλά με την πίεση του χρόνου δεν μπορούσα να τα πω όλα. Εγώ αναφέρθηκα ε, στον Μεσογειακό κόμβο, ενεργειακό κόμβο. Ε, ξέρουμε ότι υπάρχει το κοίτασμα της Αφροδίτης, είναι νέα οικόπεδα τα οποία έχουν, τη δυνατότητα μεγάλης παραγωγής όσον αφορά το αέριο οπωσδήποτε θα πρέπει να γίνει μεγαλύτερη έρευνα και ενδεχομένως να βρεθούν μεγαλύτερα αποθέματα. Ε, ε, υπάρχουν βεβαίως προβλήματα για χώρες, δύσκολη κατάσταση για χώρες όπως ε, η Κύπρος ή η Μάλτα έτσι ώστε να ξεπεράσουν αυτό το πρόβλημα που έχουν ως νησίδες ενέργειας. Θα πρέπει να δείξουμε αλληλεγγύη η οποία να φανεί και στον κατάλογο των προγραμμάτων κοινού ενδιαφέροντος που θα πρέπει να έχουμε όσον αφορά το ξεκλείδωμα αυτών των νησίδων αλυσίδων ενέργειας ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται και θα συνεργαστεί με την ε, Κυπριακή κυβέρνηση έτσι ώστε να ερευνηθεί περαιτέρω το οικόπεδο Αφροδίτη και να ε, ε, ε, ε, βεβαιωθούμε ότι η Κύπρος θα συνδεθεί με τον, με τον ενεργειακό κόμβο της Ευρώπης και θα περιμένουμε καινούριε αποκαλύψεις, ανακαλύψεις και καινούρια μεγαλύτερη συμμετοχή και της Κύπρου σε αυτήν την μικρότερη εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από εξωτερικές πηγές. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Εγώ εδώ είμαι κύριε Σεφκοβίτσα. Ε, όσον αφορά τις παγκόσμιες διαπραγματεύσεις ε, για το κλίμα. Ε, παραμένει ασαφές ένα συγκεκριμένο απλό ερώτημα. Ποιος θα διαπραγματευθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε αυτές τις διεθνείς διαπραγματεύσεις για το κλίμα. Ένα όνομα χρειαζόμαστε έτσι ώστε να ξέρουμε ποια θα είναι αυτή η φωνή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, όσον αφορά το περιεχόμενο, είπατε επανειλημμένα ότι θέλετε να είναι ουσιώδης η ε, ε, διεθνής εξέλιξη. Τι εννοείται ουσιώδης. Ε, τι σημαίνει για την Ευρώπη. Η Ευρώπη θέλει ένα, ε, ε, θέλει, έχει πιθανότητα 40% έτσι ώστε να επιτύχει το, το στόχο της, αλλά θα πρέπει να δούμε αν και οι υπόλοιπες συνθήκες είναι αυτές και έτσι ώστε να ξέρουμε ότι το μείον 40 είναι όντως μείον 40 και όχι μείον 50. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Κοιτάξτε, εάν το πρόβλημα είναι ποιο θα πάει στο Παρίσι, εγώ θα πάω στο Παρίσι. Αλλά είναι μακρύς ο δρόμος που οδηγεί στο Παρίσι ε, και ξεκινάει ήδη από την Τρίτη στις Βρυξέλλες και μετά θα συνεχιστεί στη Λίμα και μετά θα υπάρξουν και άλλες πολλές διεθνείς διασκέψεις και συναντήσεις και διαπραγματεύσεις. Επομένως, σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κάνει κανείς ε, είναι ε, να δείξει αποφασιστικότητα και ε, πνεύμα ρωμαλαίων. Γιατί το θέμα δεν αφορά μονάχα τον Αντιπρόεδρο για την Ένωση της Ενέργειας, αλλά όλοι αυτοί οι συνάδελφοι που σας έδειξε προηγουμένως στο οργανόγραμμα είναι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με θέματα τα οποία συνδέονται και με την Ενεργειακή Ένωση αλλά και με την ε, εν επιτυχία στο Παρίσι αυτό που θα ήταν το πιο αποτελεσματικό και η καλύτερη αντιπροσώπευση στις διαπραγματεύσεις αυτές είναι ε, η καλή εκπροσώπηση της ε, Κομισιόν και αυτό δεν αφορά μονάχα το αν θα πάει ο αντιπρόεδρος ε, ο οποίος ασχολείται με θέματα ενεργειακής ένωσης. Το θέμα είναι να έχουμε επιτυχία, να επιτύχουμε διεθνή νομικά δεσμευτική συμφωνία στο Παρίσι γιατί το κλίμα είναι ε, εξαιρετικά σημαντικό και για τους πολίτες και πρέπει ε, να είμαστε σίγουροι ότι και οι πολίτες θα είναι ικανοποιημένοι αλλά και η βιομηχανία δεν θα οπισθοδρομήσει. Ε, όσον αφορά το επίπεδο των ε, ε, φιλοδοξιών, οπωσδήποτε την Τρίτη θα ξέρουμε κάτι παραπάνω μετά από την έγκριση του πλαισίου για το 2030. Ωστόσο, σας λέω από τώρα ότι η προετοιμασία της Κομισιόν θα είναι πολύ φιλόδοξη όσον αφορά το Παρίσι. Ευχαριστώ θα ολοκληρώσαμε τον ε, κύκλο των, πολιτικό των εκπροσώπων των πολιτικών ε, ομάδων. Ο συνάδελφος Πίτερ Λίζε τώρα. Ναι κύριε υποψήφια αντιπρόεδρε, κύριε πρόεδρε, αναφερθήκατε στο θέμα της ενεργειακής αποδοτικότητας. Ο Ζαν Κλοντ Γιούγκερ και ο Μικέλα Αρίας Κανιέτε ήταν πολύ ακριβείς ως προς το ερώτημα αυτό. Δηλαδή 30% ε, δέσμευσης μέχρι το 2030 και θα ήθελα να μου το πείτε και εσείς με ακρίβεια και το πώς ε, μπορείτε πραγματικά να υποστηρίξετε αυτούς τους δύο να εφαρμόσουν αυτή τη δέσμευση. Το θέμα των κονδυλίων είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχει η οδηγία eco-design ε, και παρόλο που είναι λογική ως προς τον πυρήνα της, ωστόσο έχουν εκφραστεί και κάποιες κριτικές. Ε, ε, ερώτημα. Τι θεωρείτε για την ε, ρύθμιση των ντους όσον αφορά την οδηγία είπε ο κύριος Κανιέτε ότι θέλει να την συνεχίσει. Αλλά πώς θέλετε εσείς να αφαιρέσετε το κομμάτι της γραφειοκρατίας και να δώσετε ρεθίσματα ούτως ώστε να υπάρξει υποστήριξη ευχαριστώ πολύ, κύριε Λίζε. Ε, ε βεβαίως όπως είπε ο, ο πρόεδρος κ. Ε, Γιούγκερ και ο συνάδελφος Μικέλ και εγώ έχω αναλάβει αυτή τη δέσμευση του 25% στον αφορά την ενεργειακή αποδοτικότητα και θα κάνω ό,τι μπορώ ήδη αύριο στο Λουξεμβούργο. Και μπορώ να σας πω ότι όταν προετοιμαζόμουν για τη σημερινή ακρόαση αλλά και για τις αυριανές διαπραγματεύσεις με τους ε, υπουργούς ε, τα θέματα αυτά θα είναι εξαιρετικά δύσκολα στη διαπραγμάτευση ε, γιατί θα υπάρξει μεγάλη αντίσταση, αντιπολίτευση από τις χώρες μέλη. Αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ πραγματικά στη διαπραγματεύση αύριο για να εξηγήσω πόσο σημαντική είναι αυτή η στόχη για το μέλλον ε, της πράσινης πολιτικής στην Ευρώπη. Όσον αφορά το eco-design, εδώ ε, νομίζω ότι η Επιτροπή, το σύνολο της Επιτροπής θα χρειαζόταν τη βοήθειά σας όσον αφορά μια καλύτερη επικοινωνία. Ε, η οδηγία αυτή ε, έχει περιγραφεί στον τύπο και περιγράφεται σαν ένα γραφειοκρατικό εργαλείο μέσω της οποίας η Επιτροπή προτίθεται να ρυθμίσει τα πάντα από τις μικρές στους μεγάλες αφαρμογές και λησμονούμε να πούμε ότι χάρη σε αυτή την οδηγία το 2020 η Ευρώπη πρόκειται να εξοικονομήσει ένα ποσό το οποίο αντιστοιχεί στην ε, κατανάλωση ενέργειας στην Ιταλία για ένα χρόνο. Τόσο σημαντικός είναι αυτός ο στόχος και γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει απλώς να έχουμε μια καλύτερη επικοινωνία προς τα έξω. Ε, όσον αφορά τις ηλεκτρικές κούπες, προτάσεις όπως αυτή. Θα πρέπει να εξηγήσουμε στους πολίτες γιατί το προτείνουμε, ποια θα είναι τα συγκεκριμένα ωφέλη και να αποφύγουμε αυτή τη γραφειοκρατία στην οποία αναφερθήκατε. Και συμφωνώ μαζί σας, θα πρέπει να μειωθεί. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε εκείνες τις εφαρμογές που πραγματικά μπορούν να οδηγήσουν σε μια ουσιαστική εξοικονόμηση ενέργειας. Ευχαριστούμε πολύ ο κύριος Ματίας Κρότε. Ευχαριστώ πολύ, εδώ είμαι. Όταν πήραμε τα χαρτοφυλάκια για την νέα επιτροπή και ανακαλύψαμε εκεί το θέμα της Ενεργειακής Ένωσης και το γεγονός ότι το κλίμα συνδέεται με την ενέργεια ε, υπήρξαν πολλές επιφυλάξεις από τους συναδέλφους ότι τα επόμενα πέντε χρόνια το θέμα της κλιματικής πολιτικής αλλά και το θέμα της περιβαλλοντικής πολιτικής τελικά ε, θα μπει στην ε, άκρη θα παραμεληθεί. Ε, τι σκέφτεστε εσείς ως αντιπρόεδρος να κάνετε για αυτό το τομέα, γιατί οι φωνές της ε, κριτικής ε, μετριάζονται. Ε, αναφερθήκατε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είπατε κάποια συγκεκριμένα πράγματα, αλλά τι πιστεύετε ε, για το θέμα αυτό και σε σχέση με την κοινή γνώμη, γιατί υπάρχουν πάρα πολλέ υπογραφές από πολίτες. Τι θα γίνει με το περιβάλλον, αυτό είναι το ερώτημα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γκρότε για αυτό το ερώτημα. Ε, καταρχήν δεν ε, πιστεύω ότι αυτή η πολύ σημαντική περιβαλλοντική πολιτική ε, θα μπει στην άκρη. Γιατί ε, ε ξέρω πώς σας ενδιαφέρουν οι πολιτικές αυτές και μπορώ να σας διαβεβαιώσω και αυτό αναγράφεται και στο Mission Letter ε, ε, σε, μένα στον, ε, προς τον Επίτροπο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής αναφέρονται οι στόχοι αυτοί, οι προτεραιότητες αυτές και αναφέρεται πόσο σημαντικές είναι οι πολιτικές αυτές για το μέλλον. Βεβαίως θα υπάρξουν σημαντικές εξελίξεις τα επόμενα χρόνια. Όσον αφορά τις ανανόσιμες πηγές ενέργειας, υπάρχει τρίτη... Υπάρχει τρίτη, μια τρίτη πηγή παραγωγής ενέργειας. Αλλά πολύ συχνά η ευρεία χρήση σε ε, είναι περιορισμένη γιατί ε, δυστυχώς ε, δεν χρησιμοποιείται αυτή η μορφή ενέργειας και υπάρχουν πολλά εμπόδια στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά το ελεύθερο εμπόριο του, της ηλεκτρικής ενέργειας. Και βεβαίως θα θέλαμε να υπάρξει περισσότερη έρευνα και περισσότερα αποτελέσματα ερευνητικά, ούτως ώστε να αυξηθεί η ενεργειακή αποδοτικότητα των πηγών αυτών. Ε, και ξεκάθαρα αυτή θα είναι μία από τις βασικές προτεραιότητες της Επιτροπής γιατί όταν μιλούμε για αυτόχθονες ε, πηγές ή για ανεργιακή ανεξαρτησία στην Ευρώπη, αυτάρκεια μάλλον, ή για τις υποχρεώσεις που αναλάβαμε ως ε, ανεπτυγμένο μέρος ε, αυτού του κόσμου ως προς το 2015 τα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι ο παράγον κλειδί για την επίτευξη αυτού του στόχου. Ευχαριστώ. Ο Άιαν Ντόγκαν έχει το Ευχαριστώ πολύ κύριε υποψήφια αντιπρόεδρε. Θα ήθελα να σταθώ στα θέματα της ενεργειακής υποδομής. Περιμένετε να υπάρξει ανάγκη για μια νέα συνθήκη ή κάποια αλλαγή των συνδικών για να μπορέσει να υπάρξει ένα ισόπεδο γήπεδο ανταγωνισμού για τα θέματα ε, υποδομών ενέργειας. Ως ε, Σκότος ε, Ευρωβουλευτής πρέπει να σας πω ότι η Σκοτία έχει πολλές πηγές ενέργειας αλλά δεν είναι καλά διασυνδεδεμένη. Δεν μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει την αιωλική ενέργεια εάν δεν είναι πραγματικά διασυνδεδεμένος σε ένα δίκτυο. Πόσο, πότι κονδύλια λοιπόν θα χρησιμοποιήσετε, θα προσδιορίσετε ακριβώς για την ανάπτυξη αυτού του δικτύου και θα ήθελε ο λαός της Σκοτίας να ξέρει πολύ καλά αν αυτό θα βελτιώσει τις συνθήκες σύνδεσης για τα ίδια καθένα Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο κύριος Σεύτσοβιτς. Πιστεύω ειλικρινά ότι μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα με την τωρινή συνθήκη ήδη. Ξέρετε ότι είναι ακόμα πολύπλοκο το να αλλάξει η συνθήκη. Θυμόσαστε ότι η Επιτροπή Μπαρόσο 2 καθυστέρησε να αναλάβει το έργο της λόγω της διαδικασίας κύρωσης των συνθήκων. Αυτό ήταν κάτι το οποίο ήταν λοιπόν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πρέπει να εξαντλήσουμε καταρχήν το περιθώριο που έχουμε σε πολιτικό και νομικό επίπεδο με την τωρινή συνθήκη εγώ πιστεύω μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι πολλά αυτά τα οποία μπορούμε να πετύχουμε. Τώρα σε ό,τι αφορά τα προγράμματα υποδομών και τις διασυνδέσεις των ενεργειακών δικτύων. Έχουμε πολλές δυνατότητες για τη χρηματοδότησή τους. Η πρώτη δυνατότητα είναι βέβαια η διευκόλυνση Connecting Europe, Connecting Europe Facility, η οποία χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό σε επίπεδο 6 δισεκατομμύριων ευρώ περίπου. Δεν είναι τεράστιο αυτό το ποσό. Αυτό το οποίο είναι απαραίτητο να κάνουμε είναι να χρησιμοποιήσουμε καινοτόμε και δημιουργικές τεχνικές χρηματοδότησης. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις τεχνικές για να δημιουργηθούν για να φτάσουμε στα 300 δισεκατομμύρια επενδύσεων που, αν, που ανήγγειλε ο πρόεδρος Γιούνκερ. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να πετύχουμε πολύ περισσότερα. Για μένα, αυτό που είναι θετικό είναι ότι έχουμε ένα γενικό κατευθυντήριο σχέδιο για το πώς θα πετύχουμε τους ενεργειακούς μας στόχους. Έχουμε λοιπόν ένα παράτημα της στρατηγικής που αναφέρει τους συγκεκριμένους στόχους που θέλουμε να πετύχουμε το ταχύτερο δυνατό. Τα συγκεκριμένα ενεργειακά σχέδια πρέπει να περατωθούν το ταχύτερο δυνατό και αυτά που πρέπει να αντιμετωπιστούν πιο πρόθεσμα. Αν ξεκινήσουμε λοιπόν με την σωστή δημιουργία αυτού του πακέτου επενδύσεων, μπορούμε μαζί με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να προχωρήσουμε και πέραν αυτού του πακέτου για να χρηματοδοτήσουμε μελλοντικέ υποδομέ ενέργεια. Ευχαριστώ, Λέω ο πρόεδρο Μπούσεκ. Ο κύριο Χερμπράντι έχει το λόγο. Σα ευχαριστώ, κύριε πρόεδρε. <clears throat> Εδώ στο κέντρο είμαι. Κύριε Σεύτσοβιτ, σα ευχαριστώ. Αναφερθήκατε για τους πέντε πυλώνες σας, στους πέντε πυλώνες σας, την ενεργειακή απόδοση και την μείωση της χρήσης άνθρακα στην παραγωγή ενέργειας Βλέπω τις απαντήσεις σας, εσείς εστιάζετε πάρα πολύ στα ορυκτά καύσιμα και την ασφάλεια εφοδιασμού. Θα συμφωνούσατε όμως μαζί μου ότι το να είναι λιγότερο πολυδάπανη, λιγότερο βρώμικη η ενέργεια στην Ευρώπη και να εξαρτώμαστε λιγότερο από τις εξωτερικές πηγές θα πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο στις ανανεώσιμες ενέργειες και η Ανατολική Ευρώπη θα πρέπει να εστιάσει για να πετύχει το στοκοπό αυτό περισσότερο στην, στις ανανεώσιμες ενέργειες. Τώρα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα έχει μια δύσκολη διαπραγμάτευση. Ξέρουμε ότι υπάρχει μια διαίρεση μεταξύ Ανατολή και Δύσης στο Συμβούλιο. Θα μπορέσετε να πείσετε του εταίρου μα από την Ανατολική Ευρώπη ότι είναι απαραίτητο να έχουμε μια πολύ φιλόδοξη ενεργειακή και κλιματική πολιτική γιατί αυτό είναι προ το δικό του συμφέρον ήδη. Σα ευχαριστώ πολύ. Φυσικά και σίγουρα θα κάνω ήδη αύριο στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων ό,τι περνάει από το χέρι μου για το στόχο αυτό. Για μένα το πιο σημαντικό για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Πέμπτης είναι να μπορέσουμε να έχουμε σαφείς ευρωπαϊκής, ευρωπαϊκές συμφωνίες για τα θέματα αυτά. Να εξασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη κινείται όλη προς μία κατεύθυνση, έχει μία ενιαία αντιμετώπιση και έχουμε ένα κοινό πλαίσιο για να πετύχουμε όχι μόνο αυτά που είναι απαραίτητα μέχρι την συνδιάσκεψη του Παρισιού του χρόνου, αλλά μέχρι το 2020, 30 και 50. Αν δούμε τους στόχους που έχουν θεσπιστεί για το, 20, για το 2030 η Κομισιόν κάνει σαφείς αναλύσεις αντικτύπου επί τη βάση της δέσμευσή μας ότι μέχρι το 2005 ο ανεπτυγμένος κόσμος θα πρέπει να έχει μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 80 ή 90%. Με αυτό το σημείο εκκίνησης καταλήγουμε στα στοιχεία τα αριθμητικά τα οποία προτείνουμε σε εσά και στα κράτη-μέλη. Νομίζω ότι είναι όλο και περισσότερο σαφές και στις χώρες κεντροανατολικής Ευρώπης ότι είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην ανανεώσιμη ενέργεια. Υπάρχει πρόοδος, ακόμα βέβαια έχουμε διαφορετικά σημεία κίνησης για τις χώρες αυτές, διαφορετικές δυνατότητες χρηματοδότησης και διαφορετικές μορφές ε, δικτύων με διαφορετική ικανότητα να ενσωματώσουν την ανανεώσιμη ενέργεια. Πρέπει λοιπόν να έχουμε δύο στοιχεία στο πακέτο αυτό το οποίο θα συζητηθεί την Πέμπτη. Πρώτον να έχουμε μία ε, θέση από κοινού και κατανομή προσπάθειας και δεύτερον αυτό το ταμείο επενδύσεων που θα πρέπει να χρηματοδοτείται από ετήσια ε, χρηματοδότηση από το σύστημα εμπορίας εκπομπών ώστε να μπορέσουν οι ενεργειακοί σταθμοί, η παραγωγή ενέργειας να ε, ανανεωθεί και να είναι πιο καθαρή και πιο αποδοτική από ό,τι είναι σήμερα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Στις γραπτές σας απαντήσεις, κύριε Επιτροπέ, ε, ε, ε, είπατε ότι όλα τα κράτη-μέλη αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχουν πληροφορίες σωστές όσον αφορά τις διεθνείς διαπραγματεύσεις και να καταλαβαίνουν ότι είναι ενωτική και ενιαία η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις πάλι σε διεθνές επίπεδο και ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να μειώσει τις ε, εκπομπές, αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα, ε, και άλλα προβλήματα. Υπάρχουν ε, μολυντές μεγάλοι, όπως είναι ας πούμε οι Ηνωμένες Πολιτείες ή η Κίνα. Τι μπορείτε να κάνετε για χώρες οι οποίες δεν συμμετέχουν σε αυτόν τον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής. Μπορείτε να βελτιώσετε επίσης ε, την κατάσταση όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Ε, έχω την ε, δυνατότητα να μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα. Ε, μπορούμε οι δυο μας να άνετα και οι διερμηνείς θα μεταφράσουν την απάντησή μου στα σλοβακικά. Όσον αφορά τώρα το ερώτημά σας, μπορώ να σας υπασχεθώ εκ μέρους της Επιτροπής αλλά και σαν δική μου προσωπική δέσμευση ότι θα προετοιμάσουμε αυτές τις διαπραγματεύσεις ότι θα έχουν ε, μεγάλο βαθμό, υψηλό βαθμό διαφάνειας και θα ενημερωθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις διαπραγματευτικές θέσεις γιατί γνωρίζουμε ότι τα θέματα αυτά είναι πολύ σημαντικά για το Κοινοβούλιο. Μετά τη τελευταία Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών είμαι πολύ πιο αισιόδοξο όσον αφορά τους στόχους για το Παρίσι. Νομίζω ότι θα πετύχουμε πολύ περισσότερα πράγματα στο Παρίσι από ό,τι είχαμε θεωρήσει αρχικά. Ε, στη Νέα Υόρκη ε, βιώσαμε κάτι εντελώς διαφορετικό, δηλαδή μια μεγαλύτερη δέσμευση για τους κλιματικούς στόχους και ε, Είδα ότι ο Γενικός Γραμματέας, ο κ. Μπαν Κιμούν, ε, πραγματικά είναι επίσης πρόθυμος να δεσμευτεί στην κατεύθυνση αυτή. Και οι Ηνωμένε Πολιτείε ψήφισαν μια νέα νομοθεσία για τους σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ η Κίνα ε, αυτή τη στιγμή δοκιμάζει ένα καινούριο σύστημα το οποίο μοιάζει με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας των ε, Ρήπων των εκπομπών αερίων και όλα αυτά προτίθεμα να τα αξιοποιήσω την Πέμπτη ούτως ώστε να ενισχύσω την ε, διαπραγματευτική μας ε, θέση για την άνοιξη του προσεχούς ε, έτους και έτσι λοιπόν πιστεύω ότι έχουμε περισσότερα ατού στα χέρια μας και υπάρχουν πολλές πιθανότητες να λάβουν μέρος στα περισσότερα κράτη. Ο κύριος Γιάννη Γιάντος, ευχαριστώ πολύ. Κύριε υποψήφι, εδώ βρίσκομαι, στα αριστερά σας. Μας είπατε και ε, άλλωστε αφορά και την ε, επιστολή που περιγράφει την θέση σας ε, του ε, ε, πρόεδρο Γιούγκερ ότι ε, θα επιτύχετε τους καλύτερους στόχους. Πιστεύετε όσον αφορά τις ανανεώσιμες, το 27% που έχει αναφέρει ως στόχο η παλιά Επιτροπή και είσαστε μέλος του παλαιού ε, κολεγίου των Επιτρόπων και επομένως ψηφίσατε και εσείς τα μέτρα. Πιστεύετε ότι με το 27% η Ευρώπη θα μειώσει τελικά κατά 50% την ικανότητά της όσον αφορά παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή θα γίνει με λιγότερη ε, ε, προσπάθεια σε αυτή τη δεκαετία από τη δεκαετία 20-30. Πιστεύετε ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει ε, πρωταγωνιστής παριθμόν ένα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Απάντηση είναι θεμητή η ερώτησή σας. Θα σας εξηγήσω ποια είναι, αυτή, ποια είναι η λογική της προτάσεως που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το σημείο κίνηση στην αρχή ήταν πώς μπορούμε να καλύψουμε τις δεσμεύσεις μας ε, όσον αφορά τον στόχο της μείωσης της χρήσης άνθρακα ε, για το 2030 και πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό ε, με τον πιο λογικό από οικονομικής απόψεως τρόπο. Αυτή ήταν, αυτή το σημείο κίνηση της ανάλυσης και προσπαθήσαμε να βρούμε μεθοδολογικά πώς μπορούμε να φτάσουμε στο αποτέλεσμα αυτό. Ε, ε, ελάβαμε υπόψη κάποιες βασικές παραμέτρους τις οποίες σας παρουσίασα ε, και που τα κράτη-μέλη συμφώνησαν με αυτό το μείον 40 όσον αφορά την μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και είπαμε τουλάχιστον 27% όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας γιατί αυτό θα ήταν ο πιο σωστός από απόψη απόδοσης τρόπος. Θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε πιο γρήγορα αλλά το κόστος θα ήταν πάρα πολύ ψηλότερο και επομένως κάναμε και μια οικονομική ανάλυση ταυτόχρονα έτσι ώστε ε, να προτείνουμε κάτι και σε εσά και στα κράτη-μέλη που θα ήταν πιο λογικό από οικονομική απόψεως. Μπορώ να σας πω ότι ήδη τώρα είμαι πεπισμένο ότι θα ε, ξεπεράσουμε αυτό το στόχο του 27% γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές χώρες οι οποίες είναι διατεθειμένες να ξεπεράσουν αυτό το στόχο του 27%. Πιστεύω δε ότι και κατά την άποψη αυτή τελικά ε, η Ευρώπη θα ε, επιτύχει τον στόχο αυτό και θα τον ξεπεράσει. Και αυτό προς όφελος ε, των προσπαθειών μας για την κλιματική αλλαγή και κυρίως όσον αφορά τον στόχο για την μείωση άνθρακα. Jean-Luc Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Καλησπέρα σας υπογραμμίσατε τις, οικονο, ε, τις οικονομίες ενέργειας, αναφερθήκατε ε, στα 300 δις ε, τα οποία ανέφερε ο πρόεδρος Γιούγκερ και τα υποσχέθηκε σε πολλούς επιτρόπους χωρίς να ξέρουμε όμως αν υπάρχουν αυτά τα 300 δις και από πού προέρχονται. Έχω να σας κάνω λοιπόν μία πρόταση. Με τον Φίλιπ Μαϊστάχτη και τον Εμμανουέλ Μακρόν είχαμε σχεδιάσει ένα σχέδιο που θα ενέπλεκε τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία όσον αφορά την ε, ε, αποταμίευση ενέργειας καθώς επίσης και τις επενδύσεις ε, και που θα αφορούσε 350 δις. Δηλαδή στην ουσία εμείς προτείναμε από τη μία μεριά να υπάρχει η νομισματική δημιουργία η οποία να μην χρησιμοποιείται μονάχα και να μην οφείλει μονάχα τις τράπεζες αλλά τελικά ε, να δημιουργεί και καλύτερη ενέργεια. Ε, συμφωνείτε με κάτι, θα το στηρίζατε. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρότασή σας. Βεβαίως αυτό είναι ένα πολύ ευρύτερο ζήτημα το οποίο αφορά και την ε, σταθερότητα και την ανάπτυξη. Καταλαβαίνετε αυτά τα χρήματα αναφέρονται σε ένα πολύ ευρύτερο πακέτο. Και όλα αυτά βεβαίως ακόμα βρίσκονται υπό το ζήτημα είναι να δούμε πώς θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι οποιοδήποτε, οποιοδήποτε πρόγραμμα θα είναι αξιόπιστο όσον αφορά τη σταθερότητα και την ανάπτυξη και από την άλλη πλευρά θα αφορά την πραγματική οικονομία όπως είπατε και εσείς. Κατά αυτήν την έννοια βεβαίως ε, η πρόταση που κάνετε ε, όσον αφορά την ε, Τράπεζα Επενδύσεων θα μπορούσε να είναι πολύ χρήσιμη. Στην Επιτροπή Μπαρόζο 1 υπήρχε, έγινε αναφορά στα λεγόμενα ομόλογα έργου. Βεβαίως ξέρουμε ότι θα πρέπει κανείς να δει τον τρόπο με τον οποίο τα πράγματα μπορούν να λειτουργήσουν καλύτερα γιατί διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε τελικά να παράγουμε αυτά τα 300 δις και για να είμαι ειλικρινής θα πρέπει να ε, έχουμε μια Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων η οποία να είναι πιο δυναμική και η οποία να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες ε, ε, έτσι ώστε να μην ασχοληθούν μονάχα θα, θα πρέπει όλοι όσοι συμμετέχουν στις διαδικασίες αυτές να βρουν λύσεις έτσι ώστε να μπορέσουμε να συνδυάσουμε τα διαρθρωτικά ταμεία, τα ευρωπαϊκά ταμεία γενικά με επενδύσεις ε, που θα αφορούν προγράμματα δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Θα πρέπει να ε, συμμετάσχουν ε, και τράπεζες αποταμιευτικές και ταμεία τα οποία αφορούν συντάξεις, ασφαλίσεις κτλ. έτσι ώστε να φτάσουμε. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Αντώνιο Ταγιάννη. Σας ευχαριστώ. Κύριε Αντιπρόεδρε Εύκοβιτς. Ξέρουμε ότι εσείς πάντα αγωνιστήκατε για μια βιομηχανική πολιτική η οποία θα ελάμβανε ε, υπόψη το κόστος της ενέργειας καθώς επίσης και την κλιματική αλλαγή. Και βεβαίως ε, το σημαντικό ζήτημα είναι η διασύνδεση ανάμεσα στο, ε, στο πακέτο για το κλίμα του 2020 και την αποτελεσματικότητα από την άλλη για το 2030 είπαμε ότι θα πρέπει οι λύσεις από τεχνική και οικονομική άποψη να μπορούν να είναι σωστές ε, και να μπορούν να λειτουργήσουν για τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες και ότι οι βιομηχανίες οι οποίες κάνουν τη δουλειά τους καλά δεν θα πρέπει να χρειαστούν ε, να ε, υπομείνουν επιπλέον ε, ε, μέτρα τα οποία θα απεραίαν από ένα σύστημα εμπορίας ανταλλαγής εκπομπών και ένα σύστημα το οποίο θα ήταν δωρεάν και το οποίο θα τους δημιουργούσε πρόβλημα. Εσείς πιστεύετε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός έτσι ώστε να αντισταθμιστεί το κόστος του συστήματος ανταλλαγής εκπομπών. Επίσης η παραγωγή ξένη παραγωγή, παραγωγή, Κινέζοι ας πούμε, οι οποίοι ε, εξάγουν προς την Ευρώπη, πιστεύετε ότι θα πρέπει να πληρώσουν κάποιο φόρο, κάποιο δασμό ψηλότερο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ταγιάννη για τις προσπάθειές του να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ε, βιομηχανίας και για το γεγονός ότι έχει θεσπίσει στόχους για την ε, σημασία της βιομηχανίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο να φτάσει στο 20% του ΑΕΠ, του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι κέριο. Τώρα, όταν πρόκειται για το μέλλον της βιομηχανίας στην Ευρώπη, για την, ε, το ρόλο της ενέργειας στη βιομηχανία υπάρχουν δύο βασικά πράγματα. Το κόστος της ενέργειας και το κόστος του ηλεκτρισμού. Εδώ έχουμε ένα πρόβλημα. Αν δείτε το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο χονδρικής, οι τιμές είναι περίπου οι ίδιες με τις τιμές των Ηνωμένων Πολιτών. Στο επίπεδο όμως λιανικής αγοράς ενέργειας, στο επίπεδο όπου πωλείται στις επιχειρήσεις μας, η ενέργεια είναι πολύ ψηλότερη, είναι δύο ή τρεις φορές υψηλότερο το κόστος της ενέργειας. Μια αντίστοιχη κατάσταση ισχύει για το φυσικό αέριο. Δεν είναι το κόστος λοιπόν παραγωγής της ενέργειας, είναι το κόστος μεταφοράς της ενέργειας, είναι η φορολογία της ενέργειας, και εμείς ουσιαστικά μειώνουμε την ανταγωνιστικότητά μας γιατί δεν έχουμε διασυνδέσεις, δεν υπάρχει συνεργασία μεταξύ των ρυθμιστών για την ε, <clears throat> μετάδοση της ηλεκτρικής ενέργειας. Ένα άλλο σημείο που τόνισε ο κύριος Ταγιάννη είναι και αυτό πολύ εύστοχο και θα είναι και μία από τις κλίδες επιτυχίας εάν υπάρξει επιτυχία το, την Παρασκευή είναι το να εμποδίσουμε τη λεγόμενη διαρροή άνθρακο, δηλαδή τη μετεγκατάσταση επιχειρήσεων. Είναι πάρα πολύ σαφέ ότι ο μηχανισμό για την αντιμετώπιση τη διαρροή άνθρακα θα πρέπει να παραμείνει στην εργαλειοθήκη μα, <clears throat> όχι για τώρα μονάχα, αλλά και για το διάστημα επέκεινο του 2020, Αλλιώ οι επιχειρήσει μα θα μεταβούν σε άλλε χώρε όπου δεν υπάρχει σεβασμό. Ε, περιβαλλοντικής νομοθεσίας και θα έχουν τη δυνατότητα να ρηπαίνουν περισσότερο και φυσικά με τον τρόπο αυτό χάνουμε την ανταγωνιστικότητά μας και τις θέσεις απασχόλησης. Ο κ. Εντουάρ Μαρτάν έχει το λόγο. Με ναι, βεβαίως. Πολύ σωστά. Κύριε Σεφτσοβιτς, εδώ είμαι. Το χαρτοφυλάκιό σας έχει σαν τίτλο «Η Ενεργειακή Ένωση». Όπως ξέρετε και φάνηκε και με την ακρόαση της κυρίας Μπράτουσεκ, υπάρχουν πολλά ερωτηματικά για το περιεχόμενο μιας τέτοιας ένωσης. Πέραν της συνθηματολογίας, τι περιεχόμενο θα έχει αυτή η ένωση και πώς θα μας βγάλει από την τωρινή κατάσταση, γιατί αυτό είναι σημαντικό για το μέλλον της Ευρώπης. Θα ήθελα ξέρω πώς θα συνδυάσετε την εθνική, πώς θα συμβάσετε μάλλον την εθνική κυριαρχικότητα στην πολιτική ενέργεια και την αυξανόμενη σύγκληση που είναι απαραίτητη για να υπάρξει μια κοινότηση, μια ένωση στον τομέα της ενέργειας. Λέτε ότι θέλετε να έχετε ένα τρίτο πακέτο. Έτσι θα το κάνετε αυτό ή θα περιμένετε να υπάρξει ενσωμάτωση και ολοκλήρωση της αγοράς ενέργειας από τις ίδιες τις αγορές. Και πώς θα μπορέσετε να επηρεάσετε την πολιτική των κρατών μελών με ένα είδος ε, ευρωπαϊκού εξαμήνου ενέργειας. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο κ. Σεύτσοβιτς, για το ερώτημά σας. Σίγουρα θα προσπαθήσουμε να δούμε ποια θα πρέπει να είναι η τελική μορφή της Ενεργειακής Ένωσης από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Χρειαζόμαστε μια συζήτηση σε βάθος και μαζί σας και με τα κράτη-μέλη. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ για την σωστή επεξεργασία μια πρόταση για την Ενεργειακή Ένωση και θα επανέλθω ενώπιον τη επιτροπή σα για να το παρουσιάσω σε πιο λεπτομεριακό επίπεδο. Δεν νομίζω ότι το τωρινό status quo είναι αποδεκτό. Θα πρέπει να προχωρήσουμε περισσότερο και να βελτιώσουμε την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Είναι πολλά αυτά τα οποία θα πρέπει να επιτευχθούν για μια μεγαλύτερη ασφάλεια στο ενεργειακό επίπεδο και για να αναπτύξουμε καλύτερα ένα μηχανισμό αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών θα πρέπει να ξαναδούμε τα θέματα της οδηγίας για την ασφάλεια τροφοδοσίας σε φυσικό αέριο. Πρέπει να διερευνήσουμε και τις δυνατότητες να προχωρήσουμε επέκεινα του τρίτου πακέτου και πέραν των τωρινών ρυθμίσεων που ισχύουν. Γιατί θα πρέπει να έχουμε καλύτερη συνεργασία μεταξύ του υλικού και του λογισμικού ούτως υπήν σε ό,τι αφορά την υποδομή ενέργειας στην Ευρώπη. Πρέπει να έχουμε καλή αποθήκευση φυσικού αερίου, καλή διασύνδεση, αυτό είναι το υλικό αν θέλετε, καλά λειτουργούντα και ευφυή δίκτυα ενέργεια στην Ευρώπη, αλλά και το λογισμικό τη ενέργεια είναι σημαντικό. Πολλέ φορέ βλέπουμε ότι επειδή δεν υπάρχει συνεργασία μεταξύ των ε, διαχειριστών των δικτύων και επειδή έχουμε διαφορετικούς κανόνες σε εθνικό επίπεδο, διαφορετική μεθοδολογία, είναι πολύ περιορισμένο το εμπόριο ενέργειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο γιατί υπάρχει αυτή η απόκληση σε προσεγγίσεις. Πρέπει λοιπόν να αναλάβουμε την πρωτοβουλία και να εξασφαλίσουμε ότι οι διαχειριστές των συστημάτων μετάδοσης ηλεκτρισμού και οι ρυθμιστές είναι πράγματι ανεξάρτητοι και έχουν τα κίνητρα να συνεργαστούν μεταξύ τους γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να αποκομίσουμε τα πραγματικά ωφέλη μιας ενιαίας αγοράς ενέργειας. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να χρησιμοποιήσω τη δική μου γλώσσα. Γιατί φυσικά και αυτή είναι μια γλώσσα που βρίσκεται στις δικές σας γλωσσικές δεξιότητες. Κύριε Αντιπρόεδρε, εγώ ήμουν παρόν και στην ακρόαση στην Επιτροπή Μεταφορών όπου ήσασταν και εσείς παρόν την προηγούμενη εβδομάδα. Νομίζω ότι ήταν λαμπρή η παρουσίασή σας εκεί. Πιστεύω ότι και για τον τομέα της Ενεργειακής Ένωσης θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την ενεργητικότητα και την ορμή που δείξατε σε, αυτήν την, ε, σε αυτό το χαρτοφυλάκιο. Τώρα, βέβαια, η συνδίκη τη Λισαβόνα λέει ότι τα κράτη-μέλη έχουν το κυριαρχικό δικαίωμα να αποφασίσουν σε σχέση με το μείγμα ενέργεια που χρησιμοποιούν. Πώ θα μπορέσετε λοιπόν να συνδυάσετε και να συμβιβάσετε τα συμφέροντα των μεμονωμένων κρατών μελών ώστε να αποφύγουμε ένα κράτο μέλο να υφίσταται πιέσει ή να επηρεάζεται αρνητικά από τα άλλα κράτη-μέλη από την Κομισιόν. Γιατί ξέρουμε ότι όλα τα κράτη-μέλη έχουν διαφορετικέ γεωγραφικέ συνθήκες, διαφορετικά, διαφορετικές ιστορικές παραδόσεις και από αυτό μπορεί να αποκύψει μεγάλη διαφορά. Ευχαριστώ, λέει ο κύριος Σεφτσόβιτς στα Σλοβακικά. Σας ευχαριστώ για το ερώτημά σας. Φυσικά, σε ό,τι αφορά τη, στην πολιτική μεταφορών, Σας ευχαριστώ. Έχω τώρα μια νέα ε, θέση για την οποία είμαι υποψήφιο ω αντιπρόεδρο τη Κομισιόν για τα ενεργειακά θέματα. Αλλά φυσικά υπάρχει στενή σύνδεση αυτή τη πολιτική με την πολιτική μεταφορών. Θα πρέπει να τύχουν κοινού συντονισμού αυτέ οι πολιτικέ οι μεταφορέ και το διάστημα φυσικά θα πρέπει να συνδυάζονται και να συντονίζονται με την ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να βρισκόμαστε σε ένα κοινό πλαίσιο και έτσι να τα, τις αντιλαμβάνεται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για το δεύτερο σας τώρα ερώτημα, για το δεύτερο τμήμα της ερώτησής σας, μπορώ να πω ότι συμφωνώ μαζί σας. Είναι αλήθεια ότι τα κράτη-μέλη εξακολουθούν να επιμένουν ότι θα πρέπει να τηρηθεί η συνδίκη της Λισαβόνας σε ό,τι αφορά το δικαίωμά τους να προσδιορίσουν το περιεχόμενο της ενεργειακής τους πολιτικής και να παραμείνουν ανεξάρτητα και κυρίαρχα για τον προσδιορισμό του ενεργειακού μείγματος. Αλλά το ενεργειακό αυτό μείγμα μπορεί να αντιμετωπιστεί ως θέμα συζήτησης και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. είναι βέβαια βάσει τη συνθήκη στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, στην αποκλειστική αρμοδιότητα το θέμα τη ενέργεια για τα κράτη-μέλη, αλλά έχουμε ήδη μια εσωτερική αγορά και έχουμε καταφέρει να περάσουμε τρία πακέτα για τα ενεργειακά θέματα. Ω εκ τούτου, στον τομέα τη ενέργεια νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει μια καλύτερη συνεργασία και πρέπει να υπάρξει μια καλύτερη συνεργασία ώστε να εξασφαλίσουμε λοιπόν τις διασυνδέσεις οι οποίες είναι απαραίτητες και θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε γι' αυτό συμφωνίες πλαίσιο, πλαισιού. Χέλβεκ Πέτερσον. Ναι, ε, θα είμαι... Ε, ε είμαι... Not only web it's also a 360 degree hearing. Εδώ είμαι κύριε Πρόεδρε πάλι. Ε, ε χάρηκα που είπατε ότι δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ε, ότι υπάρχει αντίφαση μεταξύ της αντιμετώπισης κλιματικής ε, μεταβολής και της οικονομικής ανάπτυξης. Επίσης, ε, είπατε ότι θα ενδιαφέρεστε τόσο για την ενεργειακή ασφάλεια όσο για το θέμα της αντιμετώπισης της κλιματικής μεταβολής. Επίσης, ε, αναφερθήκατε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που θεωρώ και εγώ ότι είναι το κλειδί για τη λύση του προβλήματος. Είπατε ότι η ενεργειακή αποδοτικότητα θα πρέπει να εξεταστεί ως πρώτη πηγή ενέργειας. Το ερώτημά μου είναι πώς θα πείσετε τις χώρες μέλη ότι πράγματι ισχύει κάτι τέτοιο γιατί δεν φαίνεται να συμμερίζονται αυτή την άποψη αυτή τη στιγμή. Παρακαλώ πείτε μας κάποια πράγματα σχετικά με αυτό. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την ερώτηση. Ε, πιστεύω πράγματι ότι το επιχείρημα εδώ είναι πολύ απλό. Ε, μπορούμε να δαπανίσουμε το 46% της ε, ενέργειας, ε, του λογαριασμού της ενέργειας για την θέρμανση και τη ψήξη των κτηρίων μας δεν είναι υπερβολικά δαπανηρό όταν πληρώνουμε 400 δις ευρώ το χρόνο για την ενέργεια ε, πώς μπορούμε λοιπόν να αυξήσουμε την αποδοτικότητα στα κτίρια μας. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Όταν ε, μελέτησα τις πολιτικές αυτές και επίσης ε, ρώτησα τους συναδέλφους και τους εμπειρογνώμονες στην Επιτροπή γιατί είναι τόσο δύσκολο να πείσουμε τις χώρες μέλη και δεν μπορούμε να σημειώσουμε καμία πρόοδο ε, γιατί κατά μέ η επιλογή είναι πολύ προφανής, εξόθαλμη. Μια από τις απαντήσεις ε, που νομίζω ε, δείχνει προς σωστή κατεύθυνση είναι το ότι μέχρι τώρα είχαμε υπερβολικά πολλές ρυθμίσεις και η αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας των, κτηρίων θεωρείται μια υποχρέωση και ήταν ένα περιοριστικό, ρυθμιστικό πλαίσιο αυτό το οποίο κυριαρχούσε εδώ. Ίσως θα έπρεπε να σκεφτούμε περισσότερο ε, στην κατεύθυνση της παροχής κινήτρων. Δηλαδή πολίτες που θέλουν να έχουν μια πιο αποτελεσματική θέρμανση, ένα πιο αποτελεσματικό σύστημα θέρμανσης στα νοικοκυριά τους. Γιατί ε, έχουμε καλά μοντέλα στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες όσον αφορά την παροχή κινήτρων προς τους Δήμους και τις κοινότητες για να αντιμετωπίσουν αυτό το θέμα της αύξησης ενεργειακής αποδοτικότητας των κτηρίων ούτως ώστε οι χώρες μέλη πραγματικά να πάρουν πιο σοβαρά αυτές τις πολιτικές. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Σακοράφα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υποψήφια Αντιπρόεδρε, μια ακόμη επίπτωση της νεοφιλελεύθερης πολιτικής σας είναι η δημιουργία μιας νέας κατηγορίας κοινωνικής κατηγορίας, αυτής των ευάλωτων καταναλωτών στον τομέα της ενέργειας, οι οποίοι πλήττονται από μια νέα και πρωτόγνωρη μορφή φτώχεια την ενεργειακή φτώχεια. Γνωρίζετε την έννοια της ενεργειακής φτώχειας. Αδυναμία στοιχειώδους πρόσβαση στι απαραίτητες μορφές ενέργειας που εξασφαλίζουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο ζωής. Και μιλώ για το αυτονόητο. Πρόσβαση στο φωτισμό, τη θέρμανση, στην ψήξη δηλαδή στις ελάχιστες παροχές που θα έπρεπε να παρέχονται σε όλους αδιακρίτως, αλλά εσείς τις αντιμετωπίζετε σαν εμπορεύματα. Ερωτώ λοιπόν και θα σας παρακαλούσα για συγκεκριμένη απάντηση. Η περιβόητη ενεργειακή ένωση που φιλοδοξείται να επιτύχετε με την ιδιότητα του Αντιπροέδρου. Έχει τελικά χώρο για αυτή την κοινωνική τάξη ενεργειακής φτώχειας. Και αν ναι, πώς σκοπεύετε να κάνετε πράξη την, κοινωνική, την κοινωτική αλληλεγγύη. Συγκεκριμένα, με ποιον ακριβώς τρόπο ποια χρηματοδοτικά εργαλεία, τι ύψος πόρων και πόσο άμεσα σκοπεύετε να υιοθετήσετε και να τα διαθέσετε για να προστατεύσετε τους ευάλωτους καταναλωτές από την άνοδο των τιμών και από τους που τους οδηγεί στην ενεργειακή φτωχοποίηση. Ευχαριστώ. Thank you very much, madam. Ευχαριστώ πολύ κυρία μου για αυτή την ερώτηση γιατί πραγματικά είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Και νομίζω ότι το θέμα αυτό έχει χειροτερέψει το ζήτημα αυτό λόγω της ε, κρίσης και υπάρχει πάνω από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι που είναι στερημένοι από την, ε, που θερούνται και το ηλεκτρικό ρεύμα. Και αν σκεφτούμε τα προβλήματα του αναπτυσσόμενου κόσμου θα πρέπει να πούμε ότι λόγω ακριβώς της πρόσφατης ε, κρίσης υπάρχει και περισσότερη ενεργειακή φτώχεια και στην Ευρώπη. Ε, μας ρωτάτε τι, τι, θέλουμε να κάνουμε. Ε, ξέρετε ότι όταν το θέμα είναι κοινωνική πολιτική, αυτό, η κοινωνική πολιτική είναι πάρα πολύ στις χώρες μέλη. Ε, από, στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Βεβαίως ε, μπορούμε να διδαχθούμε ημένα από τους δε ε, όσον αφορά τη χάραξη μιας κοινωνικής πολιτικής για τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά και τους πιο ευάλωτους πολίτες. Υπάρχουν διάφορα ε, μοντέλα στις χώρες μέλη και θα μπορούσαμε να αναλύσουμε ποιο είναι το πιο ενδεδειγμένο μοντέλο για ποια χώρα. Ε, σε ορισμένε περιπτώσει άμεσα είναι για τι ευάλωτε ομάδε ε, πληθυσμού. Σε άλλε περιπτώσει οικονομική υποστήριξη για αυτού που δεν μπορούν να πληρώσουν το ηλεκτρικό. Ε, σε άλλες χώρες υπάρχουν ε, κατόφλια όσον αφορά τις βασικές ανάγκες ενέργειας για τις πιο ευάλωτες ομάδες και πάλι του πληθυσμού. Όλα αυτά είναι μοντέλα ε, που θα μπορούσαμε να αναλύσουμε συνεργασία με τις χώρες μέλη θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε τα, το κοινωνικό ταμείο, τα διαρθρωτικά ταμεία κλπ. Και είναι σημαντικό επίση να υπάρξουν ε, ε, κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τι κρατικέ ενισχύσει, γιατί θα μπορούσε αυτό να βοηθήσει ανθρώπου που βρίσκονται σε άμεση ανάγκη και οι οποίοι βεβαίω θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια σε προσιτέ τιμέ. Ε, κυρία Έγκστρομ. Ευχαριστώ πολύ κύριε υποψήφια την πρόεδρε Σεύκοβιτς. Ε, θα ασχοληθώ με το ίδιο θέμα η κλιματική στόχοι είναι πολύ καλή. Θα πρέπει να αυξήσουμε τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας και να μειώσουμε ε, το ε, κάρβουνο. Αλλά σε μερικές χώρες ε, είναι πάρα πολύ δύσκολη η επένδυση σε ανανεώσιμες. Την προηγούμενη εβδομάδα πάλι ακούσαμε ότι τα ορυκτά καύσιμα θα έχουν περισσότερες επιδοτήσεις από, τα, από τις ανανεώσιμες πηγές. Ωστόσο γνωρίζουμε ότι η ενεργειακή φτώχεια είναι ένα πρόβλημα το οποίο μεγαλώνει όλο και περισσότερο και πρέπει να αναλάβουμε δράση. Πώς θα διασφαλίσετε ότι ε, τα μέτρα για την ανάπτυξη των ε, εναλλακτικών μορφών ενέργειας θα αντιμετωπίσουν και την ενεργειακή φτώχεια. Ε, δύσκολο το ζήτημα και όχι απλή απάντηση. Αυτά είναι σημαντικές προκλήσεις ε, και για τα κράτη-μέλη και για την Κομισιόν αλλά και για την Ένωση ε, όσον αφορά το μέλλον. Το πρώτο σκέλος της απάντησής μου θα είναι το εξής, ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να ολοκληρώσουμε την ενιαία αγορά ενέργειας, ε, γιατί εάν δει κανείς τις τιμές χονδρικής για την ενέργεια, είναι συγκρίσιμες με αυτές ε, που βλέπουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μερικές φορές όμως ε, βλέπουμε ότι υπάρχει ε, πλεόνασμα ηλεκτρισμού στις αγορές μας αλλά δεν υπάρχουν αρκετές κοινέ προσπάθειες, δεν υπάρχουν TSOs, δεν, υπάρχουν, δεν υπάρχει συντονισμός και ρύθμιση και επομένως μονάχα με την ενιαία αγορά θα καταφέρουμε να έχουμε όλα αυτά τα ωφελήματα τα οποία θα μειώσουν προς τα κάτω, θα πιέσουν συγγνώμη προς τα κάτω τις ε, ε, τιμές ε, της, του ηλεκτρικού. Η δημόσια παρέμβαση στον τομέα της ενέργειας είναι 120-140 δις το χρόνο. Είναι πολλά χρήματα Δηλαδή γίνονται και υπάρχουν τα συστήματα ε, επιδότησης, αλλά παρόλα αυτά παραπονιέται ο κόσμος. Το κόστος είναι πάρα πολύ ψηλό. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει από τη μία να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι περιορισμοί της ε, ενιαίας αγοράς ενέργειας θα αρθούν έτσι ώστε να ωφεληθούμε πραγματικά από αυτή την νέα αγορά ενέργειας. Δεύτερον, θα πρέπει να έχουμε μια πολύ έντιμη συζήτηση όσον αφορά την δομή ε, της ενέργειας ε, ε, και της αγοράς ενέργειας και να είμαστε πάρα πολύ στην Ευρώπη και να είμαστε πάρα πολύ σαφείς όσον αφορά τις δυσκολίες οι οποίες ακριβένουν πολύ και την ενέργεια. Ευχαριστώ πολύ, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Σεύτσοβιτς. Έχετε πίσω σας μια εντυπωσιακή πορεία και έχετε μια μεγάλη εμπειρία για τα εξωτερικά θέματα ως διπλωμάτης. Θα ήθελα να σας παραπέμψω στο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων της Μόσχας. Η κυρία και αυτή έχει ε, βρεθεί εκεί. Έχετε περάσει κι εσείς και έχετε μια μεγάλη εμπειρία για τη διαχείριση, για θέματα διαχείρισης σε υψηλό επίπεδο. Εσείς αν σας έλεγε κάποιος να γίνετε καπετάνιος σε ένα υπεροκιάνιο, θα το κάνατε αυτό με την εμπειρία σας. Και τώρα είσαστε έτοιμος εσείς να διευθύνετε την ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχετε μεγάλο ταλέντο, μπορείτε να ετοιμαστείτε σωστά για τις ακροάσεις, να απαντήσετε τα ερωτήματα αυτά. Αλλά αν ρωτιέμαι, είναι τόσο πολύπλοκο ο τομέα τη ενέργεια. Μήπω θα έπρεπε να έχετε ειδική εμπειρογνωμοσύνη σε αυτό το θέμα, δεν θα ήταν πιο τολμηρό από εσά να το αναγνωρίσετε. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο κύριο Σέρτσοβιτ. Αναγνωρίζω ότι η εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική, είναι κέρια. Και πιστεύω ότι οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κάτι μελη μας έχουν μια μεγάλη εμπειρογνωμοσύνη στα θέματα αυτά. Αυτό το οποίο χρειάζεται στον σημαντικό τομέα αυτό και στην, στον ευραλικό αυτό τομέα χρειαζόμαστε πολιτική θέληση, χρειαζόμαστε ηγετικό ρόλο, χρειαζόμαστε τις διπλωματικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για να μπορέσουν τα κράτη-μέλη μας να ξεπεράσουν την ε, περιχαρακωμένη τους κυριαρχικότητα και να προχωρήσουν σε μια ενεργειακή ε, ένωση και χρειάζεται κανείς να έχει την ικανότητα να διαπραγματεύεται με τους τόσο σημαντικούς αυτούς εταίρους και αντιπάλους όπως είναι η Ρωσία στη συγκεκριμένη περίπτωση. Χρειάζεται λοιπόν να έχει κανείς εμπειρία εξωτερικών σχέσεων για τις διαπραγματεύσεις με άλλους εταίρους. Για την ε, σφυριλάτηση μια πολιτική εναντί τη κλιματικής αλλαγής. Πιστεύετε ότι θα είχε καλής ότι υπάρχει ένας χώρος όπου υπάρχουν περισσότερα διακυβευόμενα από ότι η συνδιάσκεψη του Παρισίου για την κλιματική αλλαγή. Πιστεύω λοιπόν ότι στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση δεν εναπόκειται μόνο σε μένα και στον Επίτροπο για την κλιματική αλλαγή, αλλά είναι θέμα και για την κυρία Μογκερίνη ως εκπρόσωπο της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να διαμορφώσουμε ένα μεγαλύτερο επίπεδο προτεραιότητας για την ενεργειακή διπλωματία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να είμαι λοιπόν απόλυτα έντιμος απέναντί σας. Πιστεύω ότι μπορούμε να συνδυάσουμε τη δική μου εμπειρία και τα, τις γνώσεις μου σε επίπεδο εξωτερικών υποθέσεων με τις απαραίτητες τεχνικές ικανότητες. Είμαι σίγουρος θα με υποστηρίξουν οι υπηρεσίες μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη στο ρόλο αυτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αντιπρόεδρε, υποψήφια Αντιπρόεδρε για τις απαντήσεις σας. Ζητώ τώρα από τον συναδελφό μου, τον κύριο Λαβία, να προεδρεύσει του δευτέρου τμήματος της ακροασής μας. Και τώρα μπορούμε να συνεχίσουμε το σύστημα ping-pong με το ερώτημα της κυρίας Κιώστιγκερ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχετε πει πολλά ήδη για τις ανανεώσιμες ενέργειες, αλλά ίσως θα πρέπει να σταθούμε σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Η Κομισιόν στην οποία εσείς ήδη συμμετέχετε και θα συμμετέχετε και στο μέλλον έχει ε, υποστηρίξει τις επιδοτήσεις για το Hinkley Point, ένα σταθμό πυρηνικής ενέργειας στο, στο Βασίλειο. Γνωρίζετε ότι είναι σαφής οι συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι η δημιουργία ε, ανανεώσιμης ενέργειας πρέπει να είναι το προέχον στα, στην ευρωπαϊκή πολιτική. Για μας είναι σαφές ότι εδώ βλέπετε να είμαστε ενώπιον μιας ε, επαναφοράς της πυρηνικής ενέργειας. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο δημιουργεί μια σημαντική, μια τεράστια στρέβλωση ανταγωνισμού έναντι της πυρηνικής ενέργειας, έναντι των ανανεωσίμων ενεργειών. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω πώς θα πώς, ε, τι θέση είχατε εσείς για την απόφαση της Κομισιόν για την έγκριση αυτών των επιδοτήσεων προς το Hinkley Point. Ευχαριστώ την απάντηση παρακαλώ κύριε υποψήφια επίτροπε. Σας ευχαριστώ κύριε Ακροστήρια για το ερώτημα αυτό και αυτό αξίζει πράγματι μία διευκρίνηση. Η απόφαση για το Hinkley Point δεν αφορούσε την προτίμηση στην πυρηνική ενέργεια εναντί ανανεώσιμης ενέργειας. Ήταν μια καθαρή περίπτωση κρατικής αρρωγής. Ήταν λοιπόν μια υπόθεση την οποία είχε αναλάβει η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού. Οι Βρετανικές Αρχές παρουσίασαν ε, πιστικά επιχειρήματα για να μπορέσουν να δοθούν αυτές οι κρατικές επιδοτήσεις στο σταθμό του Hinkley Point έδωσαν σαφή στοιχεία βάσει των οποίων προκύπτει ότι θα θέλανε 7% της ε, ενέργειας να καλυφθούν από τον σταθμό του Χίνκλι Πόντ, γιατί στην αντίθετη περίπτωση θα είχαν προβλήματα στην αγορά ενέργειας, δεν θα μπορέσουν να έχουν την απαραίτητη ε, χρηματοδότηση από τις χρηματαγορές για τη δημιουργία ενός σταθμού χωρίς την κρατική επιδότηση. Ήταν μια πολύπλοκη λοιπόν διαπραγμάτευση που έγινε με τις Βρετανικές Αρχές και η Κομισιόν επέμεινε στο να, υπάρχουν, να υπάρξουν οι καλύτεροι δυνατοί όροι για τους Βρετανούς καταναλωτές και νομίζω ότι το τελικό αποτέλεσμα σε σχέση με το κόστος αυτού του εγχειρήματο οδήγησε σε χρηματοδότηση 70% από το κράτος, 30% από τους ιδιωτικούς επενδυτές με πολύ καλύτερα αποτελέσματα για τους καταναλωτές από τις αρχές των ε, διαπραγματεύσεών μας όταν παρουσιάστηκε αυτό το θέμα στην ε, υπηρεσία ανταγωνισμού. Thank Ευχαριστούμε. Και τώρα ο κύριος Πανιό. Κύριε αντι... την αντιπρόεδρε, εγώ βρισκόμαι από... εδώ, είμαι από την άλλη πλευρά. Καταρχήν θα ήθελα πραγματικά να συγχαρώ για την ενεργητικότητά σας, για την μεγάλη σας θεληματικότητα και στα εισαγωγικά σα λόγια είπε, είπατε ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για την Ενεργειακή Ένωση είπατε ότι θα έπρεπε να είχε διαμορφωθεί ήδη από πολύ καιρό μιλήσατε και τους πέντε πυλώνες ε, και ε, βεβαίως γνωρίζουμε ε, όσον αφορά τους στόχους αυτούς ε, υπάρχουν ε, προβλήματα όσον αφορά τον τρόπο υλοποίησης αυτών των στόχων. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξή. Είστε υπέρ μιας ενεργειακής ένωσης όπως αυτή που προσεγγίζει ο κύριος Ντόναλτ Τούς Τάσκ, ο νέος ε, πρόεδρος του Συμβουλίου ή πρόκειται για μια κοινή αγορά φυσικού αερίου έτσι όπως την πρότεινε ο Ζακ Ντελόρ αλλά και ο κύριος Μπούζεκ ε, εμπνεόμενος από την ε, Ένωση Άνθρακα και Χάλιβα. Ευχαριστώ πολύ και ελπίζω να κατάλαβα καλά την ερώτηση. Η αλήθεια είναι ότι έχουν υπάρξει διαφορετικά, διαφορετικές αφετηρίες που οδήγησαν στην ε, συζήτηση αυτή, στο διάλογο αυτό. Πιστεύω ότι η Ενεργειακή Ένωση ήταν ε, ένα μοντέλο ε, των φιλοευρωπαϊστών όπως ο Γέρζι Μπούζεκ και ο Ζακ Ντελόρ, στους οποίους αναφέρθηκα άλλωστε και υπέρξαν και άλλοι πολιτικοί οι οποίοι ε, είχαν προτείνει να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση και μια από τις πιο πρόσφατες προτάσεις προέλθε από τον μελλοντικό πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον κύριο Ντόναλτ Τάσκ, Τούσκ, για να το προφέρω σωστά. Αυτό το οποίο πιστεύω ότι θα συμβεί στο τέλος είναι το εξής. Θα παρουσιάσω το δικό μου πολιτικό μοντέλο που θα βασίζεται σε αυτούς τους πέντε πυλώνε. Ενδεχομένω αν τέσσερι θα τροποποιηθεί, αλλά θα ήθελα να έχουμε ένα διάλογο να σχέση με το πώ μπορούμε να πετύχουμε μια συνένεση όσον αφορά την δομή, τι πολιτικέ το ε, πλάνο δράσης, ώστε να δούμε πώς μπορούμε να αξιολογήσουμε τα επιτεύγματά μας σε, τακτικές, ε, σε τακτά χρονικά διαστήματα. Θα ήθελα να σας πω, όσον αφορά την αγορά φυσικού αερίου, όταν διατυπώνει κανείς αυτή την πρόταση, αυτό το οποίο ακούει από τους είναι το εξή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αυτό. Υπάρχουν πολύ σύνθετες ε, κανόνες περί ανταγωνισμού, ε, σύνθετοι κανόνες του ΠΟΕ. Υπάρχουν κάποιες ε, ανησυχίες ε, συστατικά θα έχουμε μια ε, διευθέτηση που θα πρέπει να προσαρμόζεται σε κάθε περίπτωση χωριστά. Ωστόσο νομίζω ότι θα πρέπει να ξεπεράσουμε αυτές τις αρχές ανησυχίες γιατί πιστεύω ότι το επιχείρημα του πόσο δαπανάμε σε ενέργειες, πόσο μεγάλος πελάτης είμαστε ε, μετράει και πραγματικά αξίζουμε καλύτερη μεταχείριση, καλύτερες τιμές και μεγαλύτερο σεβασμό και τώρα η ερώτηση του κυρίου Τεμές Μέκερ ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Σεύκοβιτς εδώ είμαι θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα της ενεργειακής αποδοτικότητας Είπατε ε, τώρα μόλις ότι είστε η υπέρ δεσμευτικών στόχων τη ενεργειακής αποδοτικότητας και δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω 100% μαζί σας. Ωστόσο είμαι κάπως απογοητευμένος ακούγοντας ε, τα αποτελέσματα της συνάντησης κορυφής. Ε, δηλαδή οι επικεφαλής των κυβερνήσεων τελικά μίλησαν όχι για δεσμευτικούς αλλά για ενδεικτικούς στόχους. Ε, νομίζω λοιπόν ότι χάσαμε την ευκαιρία. Θεωρείτε ότι τέτοια ενδεικτικοί στόχοι τελικά θα έχουν τα αποτελέσματα τα οποία επιθυμούμε. Δεύτερον, η υποστήριξη ε, των ε, επιχειρήσεων ε, θα πρέπει να υποστηριχθεί περαιτέρω. Πώς μπορείτε να το συνδυάσετε με τις πρωτογενείς επενδύσεις στον τομέα της ενεργειακής αποδοτικότητας, τη στήριξη των επιχειρήσεων. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ερώτηση βλέπω ότι έχετε μελετήσει πολύ προσεκτικά τα αποτελέσματα από τη συνάντηση κορυφής του Συμβουλίου και είναι αλήθεια ότι το σχέδιο των απορισμάτων λέει, αναφέρει ότι όσον αφορά την ενεργειακή αποδοτικότητα μιλάμε για ενδεκτικούς στόχους. Όπως σας είπα, αύριο θα ασκήσω πίεση ούτε ώστε οι στόχοι αυτοί να αποκτήσουν ένα δεσμευτικό χαρακτήρα. Αλλά ξέρετε ότι οι αποφάσει λαμβάνουν στο Συμβούλιο μέσω συνένεση και είναι πάρα πολύ δύσκολο να προβλέψουμε ποια θα είναι η τελική έκβαση. Ωστόσο, θα ήθελα να σα πω κάτι άλλο πέρα από αυτό. Δηλαδή, βασιζόμενος στην εμπειρία που έχει ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά ε, την θέσπιση αυτών των στόχων και την ε, χάραξη πολιτικών στο τομέα της πράσινης ανάπτυξης. Ε, καμία φορά είναι σημαντικότερα από τους στόχους τα συγκεκριμένα μέτρα και συγκεκριμένες πολιτικές. Επίσης τα μοντέλα παροχής κινήτρων. Και νομίζω ότι όλα αυτά τα έχουμε στα χέρια μας, στα χέρια των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Δηλαδή, ε, ε το πώς εμείς θα επεξεργαστούμε τα αποτελέσματα του Συμβουλίου και πώς θα τα μεταφράσουμε, θα τα μεταφέρουμε σε, συγκεκριμένες συγκεκριμένε πολιτικές. Νομίζω ότι είναι μια βασική προτεραιότητα της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής η προβολή του επιχειρήματος του τεράστιου κόστους και των ενεργειακών απολειών ε, που έχουμε, καθώς και το εξαιρετικά υψηλό κόστος που πρέπει να καταβάλουν οι πολίτες, για παράδειγμα, επειδή το κτίριο στο οποίο κατοικούν δεν είναι ενεργειακά αποδοτικό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Υποψήφιο Επίτροπε, στις γραπτές σας απαντήσεις είπατε, ε, αναφέρατε ε, την ε, πρόθεση άλλων μορφών πλήν των ορυκτών καυσίμων. Ίσως θα ξέρετε και από την Πρατισλάβα ότι δεν αποφασίζεται τόσο εύκολα και απλά αυτό. Αγγίζει κάποια πράγματα η Κομισιόν αλλά δεν τα προωθεί σε βάθος ερώτηση. θα βάλετε σαφείς στόχους ή θα αγγίξετε κάποια θέματα εσείς και κάποιοι άλλοι. Ε, νομίζω ότι αναφερθήκατε ε, ε, ε, εν τέλει στα βιοκαύσιμα σε σχέση με τα ε, ορυκτά καύσιμα. ναι, κοιτάξτε, εάν πάρω την έγκρισή σας ε, αυτό το ζήτημα οπωσδήποτε θα μπει στο τραπέζι του διαλόγου. Ε, εάν προσέξει κανείς και την οδηγία σχετικά με την χρήση της γης και την αλλαγή της χρήσης γης ε, θα καταλάβει ότι μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις ε, και από το Κοινοβούλιο και από τα κράτη-μέλη αλλά ότι όλοι προσπαθούν να βρουν κάποιο κοινό τόπο όσον αφορά το θέμα αυτό. Είπατε αγγίζουμε πράγματα και δεν τα κάνουμε σε βάθος. Ναι, αλλά κοιτάξτε, αυτή η γενιά των βιολογικών τροφίμων ε, και των βιολογικών ε, παραγωγών ε, που θα πρέπει να αντικατασταθούν από καλλιέργειες για βιοκαύσιμο δεν έχουν μελετηθεί ακόμα πολύ. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν επίσης και κάποιες κοινωνικές επιπτώσεις οι οποίες δεν είχαν αντιμετωπιστεί, δεν είχαν προβλεφθεί είναι γεγονός ότι μπορούμε να κινητροδοτήσουμε τους ε, ερευνητές έτσι ώστε να μελετήσουν περισσότερο την δεύτερη ε, γενιά των ε, βιοκαυσίμων γιατί όντως θα τα χρειαστούμε στο μέλλον αλλά μπορούμε, μπορώ επίσης να σας πω ότι πιστεύω ότι τα επόμενα πέντε χρόνια θα δούμε κυρίως ε, στον τομέα των μεταφορών ε, ευρύτερη χρήση εναλλακτικών ε, μορφών ενέργειας, ηλεκτρική ενέργεια κτλ. έτσι ώστε θα μπορέσουμε να μειώσουμε και την παραγωγή διοξιδίου του άνθρακος έτσι ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε και στα βιοκαύσιμα. Ευχαριστώ πολύ. Γερίστια Μπαούνσε. Καλησπέρα κύριε Σεύκοβιτς, Σεύκοβιτς, θα αριστερά σα, το θέμα της πυρηνικής ενέργειας, το οποίο αναφέρθηκε προηγουμένως, θα ήθελα, για το σταθμό της ε, Χαρόνια, ο οποίος είναι από τους παλιότερους της Ισπανίας και βρίσκεται πολύ κοντά στις κατοικημένες περιοχές, στην ε, ε, Βιτόρια Γκαστέιτς ή στο Μπιλμπάου και η οποία έχει θεωρηθεί ότι είναι ε, επικίνδυνοι όπως κάποιοι άλλοι σταθμοί που έκλεισαν στο Βέλιο. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει αυτό, η Ισπανική κυβέρνηση εξακολουθεί να υποστηρίζει την εταιρεία η οποία διαχειρίζεται αυτό το σταθμό. Καταλαβαίνω ότι αυτό είναι θέμα των κρατών μελών, αλλά η ασφάλεια των ενεργειακών σταθμών είναι δικό σας, θέμα. Θα ήθελα λοιπόν να δω αν εσείς είσαστε έτοιμος να αντιμετωπίσετε το θέμα των πεπαλαιωμένων πυρηνικών σταθμών ή όχι. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε απόλυτο δίκιο ότι το θέμα της ασφάλειας ε, το, των πυρηνικών εγκαταστάσεων το ζήτημα, ε, αυτό το ζήτημα είναι πράγματι πάρα πολύ σημαντικό και ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να συνεργαστούμε στενά με την Ισπανική κυβέρνηση στην Κομισιόν έχουμε 180 ενεργεια, πυρηνικούς ε, επιθεωρητές ε, έτσι ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι ε, οι εγκαταστάσεις λειτουργούν σωστά και με ασφάλεια και με υψηλά πρότυπα. Τα stress tests τα οποία κάναμε μετά την τραγωδία της Φουκουσίμα έδειξαν πρόσφατα αλλά και βέβαια όλη η πραγματογνωμοσύνη που έχουμε στην Κομισιόν ότι μας απασχολεί η ασφάλεια και ε, ότι ε, διασφαλίζεται αυτή η ασφάλεια εάν υπάρχουν ή σε περίπτωση που υπάρξουν οποιασδήποτε αμφιβολίες από πλευρά της Κομισιόν όσον αφορά την ασφάλεια ή την ασφαλή λειτουργία αυτών των εγκαταστάσεων τότε οπωσδήποτε θα έρθουμε σε επαφή με την Ισπανική κυβέρνηση ε, και σε έναν ανοιχτό διάλογο αλλά με στόχο ε, πούμε στην ε, Ισπανική κυβέρνηση τι πρέπει να κάνει έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια αυτών των εγκαταστάσεων. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Έριξον. Καλησπέρα κύριε Σεύκοβιτς. Από τη Σουηδία λοιπόν είμαι. Σουηδία 10 βαθμούς λέει ο μιλητής. Λοιπόν, συμφωνώ μαζί σας ότι θα πρέπει να έχουμε ε, ένωση ενέργειας ε, και ότι θα πρέπει να αναλυθούν τα απαραίτητα βήματα έτσι ώστε να το επιτύχουμε. Αλλά Ένωση Ενέργειας ε, θα πρέπει να, αυτή η ένωση θα πρέπει να βασιστεί στην αλληλεγγύη και η κατάσταση είναι δύσκολη. Ας πούμε στη χώρα μου έχουμε επενδύσει σε ε, θερμοηλεκτρικούς σταθμούς πριν από 100 χρόνια περίπου ε, και Τώρα έχουμε τη δυνατότητα για ανανεώσιμες ε, πηγές και ε, επενδύουμε και επενδύουμε πολύ και για την ενεργική αποδοτικότητα και στην ε, βιομηχανία αλλά υπάρχουν άλλες χώρες οι οποίες εξακολουθούν να χρησιμοποιούν το κάρβουνο ας πούμε, τον άνθρακα ε, τι προτίθεστε να κάνετε απάντηση παρακαλώ λέει ο πρόεδρος μικρόφωνο σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την ερώτηση. Πρώτα απ' όλα, έχετε δίκιο ότι η ελληνική και η εμπιστοσύνη, θα προσθέσω εγώ, είναι απαραίτητα στοιχεία έτσι ώστε να μπορέσουμε να οικοδομήσουμε την ε, Ενεργειακή Ένωση της Ευρώπης. Ε, είναι πολλά και δύσκολα τα προβλήματα και υπάρχουν στιγμές όπως το 2009 όπου τα προβλήματα γίνονται ακόμα πιο έντονα. Ε, επομένως εμπιστοσύνη και καλή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών έτσι ώστε ε, να μπορέσουν ε, οι χώρες να έχουν την ενέργεια, το φωτισμό, τον ηλεκτρισμό που χρειάζονται. Η Σουηδία βεβαίως ε, είναι από τους πιο καλούς μαθητές. Πρέπει να συγχαρούμε την χώρα όσον αφορά την δομή της ε, ενέργειας της και όσον αφορά την χρήση ανανεώσιμων ε, πηγών. Βεβαίως έχουν και τις γεωγραφικές συνθήκες που τους επιτρέπουν να χρησιμοποιήσουν ανανεώσιμες πηγές και το έκαναν με μεγάλη τεχνογνωσία και με μεγάλη αποφασιστικότητα. Ε, σήμερα βεβαίως πρέπει να είμαστε και ειλικρινεί και να πούμε ότι ο άνθρακας εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη πηγή ενέργειας ε, στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Περισσότερο από το 27% της ενέργειάς μας παράγεται από άνθρακα. Μετά έρχεται η πυρηνική ενέργεια και πολύ πίσω οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και επομένως έχετε δίκιο ότι περισσότερο από το 80% της ενέργειάς μας ε, δημιουργείται από το από τον άνθρακα, 44% ας πούμε της ενέργειας της Γερμανίας παράγεται από άνθρακα και λέτε τι μπορούμε να κάνουμε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ε, ε, μια νέα τεχνολογία όσον αφορά, την, ε, όσον αφορά τον άνθρακα power stations, so they are much, much... όσον αφορά την συγκράτηση και την αποθήκευση του άνθρακα θα χρησιμοποιήσουμε την τεχνογνωσία μας για αυτά σας ευχαριστώ πολύ η κυρία Βιρκούνεν Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Σέφτσοβιτς. Είπατε προηγουμένως, το είπατε κατά επανάληψη, ότι οι ευρωπαϊκές επενδύσεις ενέργειας πρέπει να εξυγχρονιστούν και να επεκταθούν για να μπορούν οι ενεργειακοί πόροι να κινούνται ελεύθερα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να ε, μπορέσουμε να εξαλείψουμε τις ενεργειακές νήσους μέσα σε εισαγωγικά. Αλλά έχουμε πολλές τέτοιες νησίδες και στο βόρειο τμήμα της Ευρώπης από όπου προέρχομαι. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια θεωρείτε τα πιο κατεπήγοντα σχέδια, τα πέντε πιο κατεπήγοντα σχέδια για την ε, ενεργειακή ε, πολιτική της Ευρώπης και πώς θα προχωρήσουν αυτά τα πέντε σχέδια κατά την άποψή σας. Ευχαριστώ πολύ γιατί αν δείτε την κατάσταση των ενεργειακών νήσων έχουμε σίγουρα ένα πρόβλημα στη, στο Βορρά, στην Φιλανδία, στα Βαλτικά κράτη όπου βλέπουμε ότι τα ηλεκτρικά δίκτυα είναι συνδεδεμένα στις πηγές του παρελθόντος. Έχουμε προβλήματα επίσης στην ε, νησιωτική ε, Ευρώπη, στη Μάλτα, στη Γύπρο, στα νησιά της Ιβηρικής Χερσόνησό μου. Πείτε ποια είναι λοιπόν τα πέντε βασικά σχέδια για το μέλλον. Θα σας έλεγα, για μένα η καλύτερη απάντηση θα είναι να δείτε τον κατάλογο των σχεδίων τα οποία έχουν προσαρτηθεί στον ε, ε, κατάλογο για την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια και από εκεί θα δείτε ότι είναι απαραίτητο να έχουμε διασυνδέσει μεταξύ Φιλανδίας και Βαλτικών χωρών και των υπολοιπών χωρών της Ευρώπης για την διανομή ηλεκτρισμού. Αυτή τη βδομάδα ή την επόμενη βδομάδα νομίζω θα ξεκινήσει ο ενεργειακός σταθμός της Κλαϊπέδας που είναι πολύ σημαντικός ως τμήμα αυτής της προσπάθειας να ξεπεραστεί αυτή η απομονωμένη ε, κατάσταση των βαλτικών και ε, σκανδιναβικών κρατών ενώ την Φιλανδία περισσότερο. Θα έλεγα λοιπόν ηλεκτρικές διασυνδέσεις μεταξύ Φιλανδίας και Βαλτικών κρατών και επίσης ενεργειακή τερματική σταθμή στην περιοχή από όπου προέρχεστε και εσείς αυτό σημαίνει ότι θα μπορέσουμε έτσι να ξεπεράσουμε την απομόνωση των περιοχών και θα βοηθήσει και τη Φιλανδία και τα βαλτικά κράτη σιγά σιγά να ενσωματωθούν πιο αποτελεσματικά στο σύνολο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ενέργειας. <coughs> Ευχαριστώ. Ο κύριος Κάλλος Ζουρίνιου. <coughs> Εδώ είμαι κύριε ε, υποψήφιε αντιπρόεδρε έχετε ένα πάρα πολύ σημαντικό καθήκον, μια σημαντική αποστολή, να μπορέσετε να βάλετε την Ευρωπαϊκή Ένωση στο επίπεδο πρωτοπόρου για την πράσινη ανάπτυξη και τις ανανεώσιμες ενέργειες και συγχρόνως να εξασφαλίσετε την ασφάλεια εφοδιασμού και την ανταγωνιστικότητα. Τρία ερωτήματα. Πρώτον, για το πακέτο ενέργειας και κλιματικής αλλαγής. Θεωρείτε ότι είναι ικανοποιητικό το 27% για τις ανανεώσιμες ενέργειες. Δεν θεωρείτε ότι το 30% θα είναι μεγαλύτερη αξιοπιστία στις δηλώσεις του Ζαν Claude ότι η Ευρώπη θέλει να είναι πρωτοπόρος και ηγέτης στις ανανεώσιμες ενέργειες. Δεύτερον για τις διασυνδέσεις έχουμε για να έχουμε πράσινη ανάπτυξη πρέπει να έχουμε καλές διασυνδέσεις ενέργειες. Πώς θα μπορέσετε να το επιτύχετε αυτό, ιδίως στην περίπτωση της ε, Ιβηρικής Χερσονήσου, η σύνδεση με την Γαλλία Τρίτον, υπάρχουν ορισμένε κυβερνήσει οι οποίε έχουν περικόψει αντί να αυξήσουν τα κίντρα για τη χρήση ε, ανανεώσιμε ενέργειε. Ποια είναι η άποψή σα για αυτέ τι πρακτικέ αυτών των κρατών Ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινήσω από το τέλος της ε, ερώτησής σα. Το πρώτο τμήμα ουσιαστικά το έχω απαντήσει ήδη. Είναι σημαντικό ότι η Πορτογαλία και η Ισπανία βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση γιατί δεν έχουν πετύχει ακόμα, είναι πολύ μακριά από το στόχο διασύνδεσης ενέργειας μεταξύ κρατών μελών. Θα θέλαμε να είναι 10% αλλά μεταξύ Πορτογαλίας, Ισπανίας και Γαλλίας είναι μόνο 2 με 4%. Είναι πολύ μικρό το ποσοστό αυτό, είναι απαράδεκτη κατάσταση. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να βρούμε καλές απαντήσεις σε αυτό το πρόβλημα. Ήδη θα πρέπει να υπάρξουν αποφάσεις την Πέμπτη και αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένα πρόβλημα προς λύση, ένα πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με σωστή χρηματοδότηση και τόσο η Ισπανία όσο και η Πορτογαλία θα πρέπει να μπορέσουν να συνδεθούν πλήρως με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο. Η Κομισιόν όπως σας είπα είναι έτοιμη να παίξει το ρόλο του έντιμου διαμεσολαβητή, όχι μόνο για αυτό το πρόβλημα αλλά και για άλλες περιπτώσεις όπου βλέπουμε ότι σε περιφερειακό επίπεδο είναι πολύ να μπορέσει να εξευρεθεί μια συνένεση. Είμαι έτοιμο λοιπόν να συμμετάσχω στι διαπραγματεύσει αυτού του είδου γιατί νομίζω ότι αυτέ οι καταστάσει θα πρέπει να ξεπεραστούν. Δεύτερο πρόβλημα που θέτεται είναι και αυτό σημαντικό. Έχουμε μια κατάσταση στην Ισπανία, την Πορτογαλία, επίση και στη Τσεχική Δημοκρατία, όπου έχουν εγκριθεί κάποια συστήματα για οικονομική υποστήριξη τη χρήση ανανεώσιμη ενέργεια. Και μετά αυτέ οι πολιτικέ έχουν αναστραφεί. Η Πορτογαλία για μένα είναι καλύτερο παράδειγμα γιατί εκεί έγινε μια διαπραγμάτευση μεταξύ της κυβέρνησης και των εκπροσώπων <clears throat> για την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας και υπήρξαν κάποιες συμβαστικές λύσεις. Σε άλλες περιπτώσεις όμως τα πράγματα έχουν εμπλακεί σε πολύπλοκες νομικές μάχες σε σχέση με την ε, με τον αναδρομικό χαρακτήρα ορισμένων αποφάσεων. Εγώ θα προτιμούσα αντί να υπάρχουν νομικές διαμάχες να γίνουν πραγματικές διαπραγματεύσεις. Κύριε Βυσνιεύσκα. Ευχαριστώ πολύ. Το θέμα είναι το εξή. Ποια είναι η δική σας ε, θέση όσον αφορά στην ε, ε, διασένεση μεταξύ ενεργειακού πακέτου και ανταγωνιστικότητας ε, ε, και εξάρτηση, συγγνώμη. υπάρχει μεγάλη εξάρτηση Ευρώπης από τη Ρωσία, η Πολωνία από την οποία εγώ προέρχομαι είναι και αυτή σε δινή θέση. Ε, εισάγουμε τα δύο ε, τρίτα του αερίου. Αλλά ωστόσο η δική μας, και η δική μας ενεργειακή παραγωγή βασίζεται στον άνθρακα. Ε, θεωρείτε ότι έχει έρθει κατάλληλη στιγμή για την χάραξη μιας ενεργειακή ε, πολιτική στην Ευρώπη που δεν αποκλεί ε, τις ε, πηγές του άνθρακα γιατί η παραγωγή ενέργειας από άνθρακα αντιμετωπίζουν μεγάλο ανταγωνισμό ε, ε, από χαμηλό, χαμηλού κόστους άνθρακα. Ευχαριστώ πολύ δεν βλέπω να υπάρχει αυτή η αντίφαση στη νέα ατζέντα ε, με τους στόχους ανταγωνιστικότητας όσον αφορά τον ε, άνθρακα ε, στην Ευρώπη. Νομίζω ότι θα πρέπει αυτά τα δύο να αναπτυχθούν παράλληλα και να ενισχυθούν αμοιβαία. Γιατί ε, όταν, όσον αφορά τα, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αυτές είναι ε, ε ντόπιε πηγές ενέργειας. Η αιωλική ενέργεια, η ηλιακή ενέργεια. Ε, με τον τρόπο αυτό γινόμαστε πιο ανεξάρτητοι από την εισαγωγή ενέργειας, εισαγωγή φυσικού αερίου από τη Ρωσία κυρίως με την οποία σε αυτή τη συγκυρία βρισκόμαστε σε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να δουλέψουμε και για τις δύο πολιτικές ταυτόχρονα και μπορούμε να πετύχουμε καλά αποτελέσματα. Όπως σας είπα, η απόφαση για το ενεργειακό μείγμα είναι μια κυρίαρχη απόφαση των χωρών μελών, αλλά ταυτόχρονα κάθε χώρα μέλος θα πρέπει να σέβεται τους κοινού στόχους στους οποίους έχουν αποδεχθεί οι χώρες μέλη. Γι' αυτό είναι σημαντικό να υπάρξει μια κοινή ευρωπαϊκή γραμμή ε, για ε, την, τις πράσινες πολιτικές και για μια πιο πράσινη στρατηγική για το μέλλον. Ε, νομίζω ότι το πακέτο 2030 θα είναι θετικό για την Πολωνία γιατί υπάρχουν δύο σημαντικά πολιτικά στοιχεία σε αυτό το πακέτο. Πρώτον, η δημιουργία Ε, η ενίσχυση μάλλον της ε, έρευνας, και ε, έρευνας για, την, για μεθόδους δέσμευσης και αποθήκευσης της ενέργειας. Επίσης σταθμή συμπαραγωγής ενέργειας ούτε ώστε και η Πολωνία να υιοθετήσει πιο φιλόδοξους στόχους στην πράσινη ατζέντα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε υποψήφιε επίτροπε, ε, σε συνέχεια των απαντήσεων σας μέχρι στιγμή, ε, θα ήθελα να πω ότι γνωρίζουμε ότι αναπόκειται στι χώρε μέλη να λάβουν τις αποφάσεις για το ενεργειακό μείγμα που θέλουν να χρησιμοποιήσουν. Η ερώτησή μου έχει ω εξή. Πώς ε, σχεδιάζεται να... προγραμματίζεται τη συνεργασία μεταξύ των χωρών όσον αφορά τι ενεργειακέ πολιτικέ, και θα ήθελα να μας πείτε κάποια πράγματα για την ε, δυνατότητα διαφοροποίησης ε, των πηγών ε, παροχής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω ότι, απάντηση, πιστεύω ότι ο καλύτερος συντονισμός και η διαφοροποίηση είναι παράγοντες κλειδιά στην δημιουργία μιας ε, ενεργειακής ένωσης στην Ευρώπη. Χωρίς καλό συντονισμό και χωρίς ε, μια διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας δεν νομίζω ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε μια Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση. Όσον αφορά το συντονισμό νομίζω ότι έχουμε ήδη μια θετική εμπειρία με τις ομάδες συντονισμού για το φυσικό αέριο και νομίζω ότι εδώ έχει, υπάρχει ένα κλίμα εμπιστοσύνη ε, και υπάρχει όλο και περισσότερη διαφάνεια στις συναντήσεις της ομάδας. Και ε, νομίζω βεβαίως ότι οι χώρες μέλη θα πρέπει να είναι έντιμες όσον αφορά τις ε, συνθήκες διαπραγμάτευσης. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει μια κοινή γραμμή στις επαφές με τις τρίτες χώρες για να εξασφαλίσουμε οι εταίροι μας να μην παίξουν στο χαρτί του Διέρη και Βασίλευε απέναντι στην Ευρώπη. Νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το πλαίσιο αυτό που ισχύει για την ε, ομάδα συντονισμού για το φυσικό αέριο και για τις άλλες πηγές ενέργειας. Τώρα, όσον αφορά τη διαφοροποίηση, το πρώτο στοιχείο κλειδί για το αέριο, ε, και έμαθα κάποια πράγματα από την αποτυχία του Ναμπούκο, ε, θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο, να έχουμε πια πιο συγκεκριμένη πολιτική παρουσία ε, σε όλες τις χώρες ε, εκεί όπου φτιάχνεται αυτός ο αγωγός του νοτίου διαδρόμου ε, Επίσης θα πρέπει να έχουμε καλύτερη επαφή με την εταιρεία που φτιάχνει αυτόν τον αγωγό ε, και θα πρέπει να υπάρχει επαρκής ε, υποστήριξη για τα έργα αυτά. Επίσης θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τα ενεργειακά τερματικά, τις νέες σχέσεις με την Αλγερία ή χώρες όπως είναι η Βραζιλία ή άλλες χώρες από τις οποίες επίσης θα μπορούσαμε να προμηθευτούμε ενέργεια εφόσον βεβαίως ε, δημιουργήσουμε τις κατάλληλες υποδομές. Hvala Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Κύριε Σεύκοβιτσε, ε, χαίρομαι, χαίρομαι που μιλάτε ε, για αυτά τα θέματα. Υπενθυμίσατε και τις ε, τους διαχωρισμούς που υπάρχουν στην Ευρώπη και ότι βεβαίως η ενέργεια δεν πρέπει πια να χρησιμοποιείται σαν πολιτικό όπλο. Μιλήσατε και για τη Ρωσία. Θα ήθελα να μου πείτε συγκεκριμένα όσον αφορά την ενέργεια. Πώς θα διαχειριστείτε πώς προτίθεστε να διαχειριστείτε τις σχέσεις με την Ρωσία, κυρίως όσον αφορά την ενεργειακή ασφάλεια. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Ξέρετε ότι επί σειρά ετών η Ρωσία ήταν στρατηγικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα η κατάσταση στην Ρωσία είναι βεβαίως πολύ στρατηγική, αλλά οι εταίροι έχουν ε, διαφορετικές θέσεις. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε σαφείς, ανοιχτοί και διάφανοι στις σχέσεις μας με τη χώρα αυτή. Και θα πρέπει σαφώς να δηλώσουμε τη θέση μας όσον αφορά την, ε, τις ε, ε, ρωσικές εταιρείες οι οποίες επιχειρούν ε, στο στην ενωσιακή επικράτεια θα πρέπει σαφώς να σεβαστούν τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι σαφές. Θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι Όσον αφορά, λέω, τον τομέα της ενέργειας θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα την ε, ε, δυνατότητα που έχει η Ευρώπη ή που πρέπει να έχει για μια συνολική αγορά. 52% ε, του, των εσόδων της Ρωσικής Ομοσπονδίας αφορά την, τα προϊόντα ε, ενέργεια. Δεν είναι δηλαδή ότι από την καλή τους καρδιά εξάγουν ενέργεια σε μας. Ε, είναι απαραίτητη αυτή η εξαγωγή για τη χώρα. Θα πρέπει να διευρύνουμε λοιπόν τη σχέση και θα πρέπει σαφώς να μπορούμε να μιλάμε με μία φωνή όπως συνέβη φέτος. Ο πρόεδρος Πούτιν έστειλε ας πούμε 18 επιστολές σε αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων αλλά η απάντηση που έλαβε ήταν μία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έτσι πρέπει να συνεχίσουμε και στο μέλλον. Ο κύριος Σεμπτάνης παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ οι απαντήσεις σας είναι πολύ ενθαρρυντικές ε, και χαίρομαι που θα συμμετάσχετε ε, στο, στη άρχιση του Παρισιού και βεβαίως ε, πολύ ενθαρρυντικές είναι και οι γραπτές απαντήσεις που μας δώσατε. πραγματικά καταλαβαίνουμε ότι θέλετε να έχετε πλήρη ρόλο στο Παρίσι. Σε σχέση με την κλιματική πολιτική, τι θα κάνετε έτσι ώστε ε, να μην ασχοληθεί μόνο με το κλίμα η συζήτηση στο Παρίσι και τι θα κάνετε έτσι ώστε ε, να ε, συνεχίσουν σωστά οι διαπραγματεύσεις και στα πλαίσια των Ηνωμένων και να καταλήξουν σε δεσμευτικές αποφάσεις. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Σας απαντώ αμέσως. Όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για την διάσκεψη του Παρισιού και την ίδια τη διάσκεψη. Όπως και σε προηγούμενες διασκέψεις βεβαίως, ξέρουμε ότι η εκπροσώπηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα είναι ε, μεγάλη, θα είναι επίσης ε, πολύ προσεκτική ε, όσον αφορά τις συζητήσεις και βεβαίως και όσον αφορά και το και βάση και του ε, της συμφωνίας πλαισίου που διαπραγματεύονται το Κοινοβούλιο με την Κομισιόν είναι σαφής, είναι ο μηχανισμός, είναι καθαρός για τον τρόπο με τον οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να πληροφορείται την ε, ε, έκβαση των διαπραγματεύσεων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και βεβαίως θα διασφαλίσω τη σωστή σας διαβούλευση και πληροφόρηση στο δρόμο προς ε, το, τη διάσημη κορυφής ε, του Παρισιού. Όσον αφορά τώρα την ενίσχυση της ε, στήριξης των πράσινων πολιτικών και των ανανεώσιμων των πολιτικών για τις ανανεώσιμες πηγές θα πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι το ζήτημα και τα κράτη-μέλη οπωσδήποτε, ότι το ζήτημα δεν αφορά μονάχα την προστασία του περιβάλλοντος, είναι και οικονομικό ζήτημα. Μας δίνει μεγαλύτερη ανεξαρτησία, μας βοηθάει όσον αφορά τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας, δημιουργεί θέσεις εργασίας. Γιατί ε, ήταν πραγματικά ε, ένας από τους λίγους τομείς που κατάφερε να κρατήσει τις θέσεις εργασίας. Επίσης ξέρουμε ότι στην Ευρώπη έχουμε αναπτύξει τεχνογνωσία, τεχνικές ε, γνώσεις καλές και είναι γεγονός ότι σε, χώρες, σε σχέση με χώρες όπως η Κίνα ας πούμε είναι γεγονός ότι η Ευρώπη έχει αναπτύξει σημαντική τεχνολογία, πράσινη τεχνολογία. Ευχαριστώ. Μαΐ Ζαν Μαρινέσκου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υποψήφια Επίτροπε, δεν θα έχουμε την ευκαιρία να δουλέψουμε για τα δύο ευρωπαϊκά δίκτυα, αλλά σίγουρα για τα θέματα της ενέργειας. Όπως ξέρετε, οι συνθήκες προβλέπουν όταν υπάρχουν δυσκολίες για την ενεργειακή παροχή, τη δυνατότητα για την Κομισιόν να προτείνει λήψη μέτρων για να λυθεί, για να αντιμετωπιστεί μια τέτοια κρίση. Εάν ανακύψει μια τέτοια κατάσταση φέτος το χειμώνα, παραδείγματος χάρη, θα χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα και τι είναι τα, ποια είναι τα μέτρα τα οποία θα προτείνετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα είμαι έτοιμο να δουλέψω μαζί σα για τα TNT, για τα TENI, τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας και η μεταφορών δεν έχει σημασία, αν σταθούμε στο θέμα του επερχόμενου χειμώνα. Εγώ πιστεύω ότι ο αντιπρόεδρος κ. Ότιγκερ θα έχει ήδη μια επιτυχία αύριο γιατί μίλησα μαζί του πρώτο έρθω σε αυτή την ακρόαση μου είπε ότι είναι δύσκολες διαπραγματεύσεις αλλά εξακολουθεί να είναι αισιόδοξο ότι μετά από τη σημερινή συνεδρίαση και τη συνέχεια που θα δοθεί αύριο στις Βρυξέλλες θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κοινό έδαφος, σε ένα κοινό πλαίσιο όπου θα καθοριστούν οι λύσεις για αυτό το χειμώνα και το επόμενο έτος. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά όχι μόνο για την Ουκρανία και τη Ρωσία αλλά και για την Ευρώπη. Πιστεύω μια σωστή λύση αυτού του προβλήματος θα καταπραίνει πάρα πολύ τι ανησυχίε οι οποίες υπάρχουν ιδίω για την αγορά ενέργειας. Τα θετικά νέα τώρα είναι ότι τα αποτελέσματα των τεστ αντοχής είναι πολύ θετικά και η Ευρώπη γενικά τα καταφέρνει πολύ καλά μπορεί να αντιμετωπίσει έξι μήνες πλήρους αποκοπής από τροφοδοσία από το ρωσικό αέριο, 5-6 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα για το φυσικό αέριο, είναι ένα ποσοστό 2-3% της κατανάλωσής μας στο φυσικό αέριο. Βέβαια για ορισμενα κάτι κράτη-μέλη μπορεί να είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση γιατί εξαρτώνται από το φυσικό αέριο της Ρωσίας πολύ περισσότερο. Αν συμβεί κάτι τέτοιο και αν βρεθούμε σε μια τέτοια έκτατη κατάσταση, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία που έχει στα θέση της και όλες τις εξουσίες της, ώστε να μην επαναληφθούν αυτά που έγιναν το 2009 και δεν θα αντιμετωπίσουμε πάλι μια κατάσταση όπου οι πολίτες στα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις στην Ευρώπη θα είναι στο σκοτάδι λόγω έλλειψης ενέργειας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Η ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης περνάει μια κέρια χρονική περίοδο που θα διαμορφώσει και το μέλλον της. και έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τους στόχους του 2030. Τα ερωτήματα μου είναι πρώτον τι συμπεραίνεται από τα τεστ αντοχής των πυρηνικών σταθμών και πώς η Κομισιό θα χρησιμοποιήσει αυτά τα αποτελέσματα και δεύτερον, ποια είναι η δική σας προσωπική αντιμετώπιση για την πυρηνική ενέργεια στην Ευρώπη. ως ένα μεταβατικό στάδιο παραγωγής ενέργειας στο δρόμο για μια οικονομία χαμηλού, χαμηλής κρίσης άνθρακος. Και δεύτερον, ποιος είναι ο ρόλος που θα πρέπει να διαδραματιστεί στην Ευρώπη, ευρωπαϊκή πολιτική, από τη γερμανική ενεργειακή πολιτική που είναι κέρια για τις χώρες κεντροανατολικής Ευρώπης. Ευχαριστώ. Εγώ πιστεύω ότι τα τεστ αντοχής <clears throat> των πυρηνικών σταθμών στην Ευρώπη έχουν παίξει ένα σημαντικό ρόλο, ήταν ιδιαίτερα σημαντικά υπό την έποψη της ασφάλειας και για να εξασφαλίσουν την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών που στο έδαφος τους υπάρχουν αυτοί οι πυρηνικοί σταθμοί ότι ανταποκρίνονται στα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμα λοιπόν αυτά τα τεστ αντοχής, ιδίως διότι μπόρεσαν έτσι να μεταλαμπαδευτούν βέλτιστες πρακτικές ούτε, ούτως ώστε οι πιο σύγχρονες, οι πιο τελευταίες εν πάση περιπτώσει, γνώσεις και εμπειρίες που έχουμε για την ασφάλεια των ποινικών σταθμών μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από άλλες χώρες. Σε 16 χώρες υπάρχουν πυρηνικοί σταθμοί, 14 από αυτές τις χώρες θέλουν να συνεχίσουν τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας, γι' αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό να δημιουργηθεί το κατάλληλο πλαίσιο ώστε όλοι οι πυρηνικοί σταθμοί οι οποίοι σέβονται τις προδιαγραφές ασφαλείας να μπορέσουν να διατηρηθούν. Στη συνέχεια έχουμε αντιμετωπίσει μία σειρά από σενάρια ώστε να μπορέσουμε να μειώσουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος μέχρι το 2050 και να έχουμε μια μείωση 80% έως 90% μέχρι το ορόσημο του 2050. Τρία από αυτά τα πέντε σενάρια που έχουν αντιμετωπιστεί και μας οδηγούν σε αυτό το στόχο συμπεριλαμβάνουν και την πυρηνική ενέργεια ως πηγή φτωχή σε εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος και αυτή τη στιγμή φυσικά είναι η δεύτερη σημαντικότερη πηγή ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να τη θεωρήσουμε ως ένα στοιχείο του ενεργειακού μείγματος που θα συνεχιστεί να είναι σημαντικό στο μέλλον, βέβαια εφόσον ανταποκρίνεται στις ε, συνδίκες ασφαλείας. Ε, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σεύκοβιτς, όταν μιλάτε για ενεργειακή αποδοτικότητα εννοείται ενεργειακή εξοικονόμηση. Τι θα κάνετε με εκείνες τις χώρες ε, μέλη που θα μπορούσαν ε, να έχουν κάποια προοπτική ανάπτυξη. Δεύτερον, είπατε ότι οι ανανεώσιμε πηγές ενέργειας μα ανήκουν. Υπάρχουν χώρε που έχουν πάνω από 30% μερίδιο. Ε, ε, θα πρέπει και αυτές να υπογραφούν σε εξοικονόμηση ή θα τις εξαιρέσετε. Τρίτον, ε, είπατε ότι ίσως τους ε, ενδεικτικούς στόχους δεν θα πρέπει να τους πάρουμε τόσο σοβαρά. Ε, σημαντικός ε, είναι ο νομοθετικός ρόλος του Κοινοβουλίου. Ε, θέλετε να έχετε μία δεσμευτική οδηγία για το Αιγαίο, για παράδειγμα, για τα ντους ε, δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να περάσει αυτό στην Σκανδιναβία και στην Αυστρία που θα πρέπει να έχουμε νέα τηλέφωνα του ντους, νέες κεφαλές, εκεί όπου δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με το νερό. Τι θα γίνει με την εφαρμογή μέτρων σε χώρες ε, για τις οποίες δεν έχουν τα μέτρα αυτά απολύτως κανένα νόημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, για το δίλημα που εκφράσατε μεταξύ ενεργειακής ε, αποδοτικότητας και βεβαίως της ε, πίεσης για ενεργειακά αποδοτικούς στόχους αλλά όταν το ζητούμενο είναι η συγκεκριμένη εφαρμογή αυτών των πολιτικών κλπ, τα πράγματα δεν είναι πολύ απλά. Βεβαίω μπορούμε να μιλάμε για ενεργική αποδοτικότητα των κτηρίων, αλλά δεύτερο σημαντικό κομμάτι για την αύξηση ενεργικής αποδοτικότητας είναι η οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό. Ε, το eco-design και αν δούμε ε, ποια είναι η εξοικονόμηση ενέργειας εδώ είναι πραγματικά εντυπωσιακά τα αποτελέσματα αλλά δεν τα αναφέρουμε συχνά ε, μέχρι το 2020 θα εξοικονομήσουμε το ίδιο ποσό ενέργειας που καταναλώνεται στην Ιταλία σε ένα έτος μόνο με την εφαρμογή της ε, οδηγίας οικολογικού σχεδιασμού. Και αυτό βεβαίως είναι ένα από τα μέτρα που δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλή και έχουν γελιοποιηθεί από τον τύπο. Αλλά θα πρέπει να αντιλήσουμε κάποια διδάγματα από εδώ. Ε, Υπάρχουν κάποιες τεχνικές ε, μελέτες για τα σεσουάρ ε, μαλλιών και για τις ε, μηχανές καφέ. Και βεβαίως εδώ δεν θα πρέπει να υπάρχουν δεσμευτικοί κανόνες γιατί στο κομμάτι αυτό η εξοικονόμηση ενέργειας δεν είναι τόσο σημαντική ώστε να πρέπει να έχουμε δεσμευτικούς κανόνες. Αλλά όταν μιλάμε για θερμοσύφωνες εδώ τα πράγματα είναι διαφορετικά, άρα θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τον οικολογικό σχεδιασμό, ούτως ώστε να πετύχουμε καλά αποτελέσματα. Ε, και εφόσον το πετύχουμε θα έρθω εδώ ε, και θα σας ε, ρωτήσω, θα ζητήσω και τις προτάσεις για το ποια είναι η καλύτερη προβολή αυτής της πολιτικής και επικοινωνία. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Μίρια Μντάλη. Ευχαριστώ πολύ κύριε υποψήφια αντιπρόεδρε Σεύκοβιτς. Είναι σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αποκτήσει ενεργειακή πολιτική η οποία να διασφαλίζει την ενεργειακή ασφάλεια αλλά και την ενεργειακή αποδοτικότητα. Ε, θα διασφαλίζει την συνέχιση των ενεργειακών πόρων ε, και θα ε, άρει τα εμπόδια αυτών των ε, πασίγνωστων νησίδων ενέργειας που έχουν πρόβλημα διασύνδεσης. Ε, κατά την άποψή σας πώς μπορούμε να ενθαρρύνουμε τις ε, επενδύσεις στις διασυνδέσεις, στις γραμμές παραγωγής, στους τερματικούς σταθμούς. Ποιο είναι το όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο θα στρέφεται προς την Ένωση Ενέργειας ενέργειας και τι θα κάνετε όσον αφορά ε, τις διασυνδέσεις ε, γιατί θα πρέπει όλοι, όλα τα κράτη-μέλη να είναι διασυνδεδεμένα με το δίκτυο του, του, της ενέργειας. Είστε από τη Μάλτα νομίζω. Είναι γεγονός ε, ότι μέχρι τώρα είναι γεγονός ότι ασχοληθήκαμε πιο πολύ με τις χώρες της Βαλτικής, τη Φιλανδία, με αυτές τις νησίδες ε, ενέργειας. Αλλά έχουμε τέτοιες νησίδες ε, και το είπα και προηγουμένως ε, και στο, στη Νότια Ευρώπη. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό γιατί είναι πρόβλημα αλλά είναι ταυτόχρονα και ευκαιρία. Αν δει κανεί ε, πώ θα πρέπει να διαφοροποιηθούν οι πηγέ ενέργεια, αν δει κανεί τι ευκαιρίε οι οποίε ε, ε, υπάρχουν όσον αφορά τη δημιουργία ενό μεσογειακού κόμβου ενέργεια, νομίζω ότι μπορεί να αποτελέσει ένα πραγματικό trading place για το φυσικό αέριο η περιοχή αυτή. Ε, μιλήσαμε προηγουμένως ε, και για τα νέα ε, κοιτάσματα φυσικού αερίου αναφερθήκαμε και στο οικόπεδο Αφροδίτη της Κύπρου όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά στοιχεία όσον αφορά την διαφοροποίηση τη στρατηγική διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας όσον αφορά τη χώρα σας γνωρίζω την ιδιαιτερότητα της και ένα πρόγραμμα προτεραιότητας ε, ε, στα θέματα και στα προγράμματα κοινών ε, και στο, στον κατάλογο των κοινών προτεραιοτήτων είναι ακριβώς ένα σχέδιο διασύνδεσης της Μάλτας έτσι ώστε η Μάλτα και η Σικελία να, ξεπεράσει, να ξεπεράσουν το, την ενεργειακή τους απομόνωση να ε, βοηθηθεί και η Μάλτα στη διασύνδεσή της με αυτόν τον ενεργειακό κόμβο. Ευχαριστώ πολύ η κυρία Γκαρντίνη. Με μικρόφωνο παρακαλούμε. Χωρίς μικρόφωνο η κυρία Γκαρντίνη. Λοιπόν, πολλά ακούσαμε όσον αφορά την ενεργειακή πολιτική και οπωσδήποτε ε, ο προβληματισμός μας γενικά αυτή την περίοδο είναι μεγάλος. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στη διάσκεψη του Παρισιού το 2015. Ε, μετά την Κοπεχάγη εγώ παρακολουθώ όλες αυτές τις διασκέψεις και πρέπει να πω ότι οι προσδοκίες που έχουν καλλιεργηθεί κάθε φορά είναι πολλές και τελικά μετά ε, βλέπουμε ότι έχουν γίνει λίγα εγώ άρχισα να ξανά να σκέφτομαι ότι αυτή τη φορά θα είναι η καλή φορά αλλά παρόλα αυτά ακούω διάφορα πράγματα εντωμεταξύ τα οποία ε, με οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ενδεχομένως δεν θα καταφέρουμε ούτε αυτή τη φορά να υπογράψουμε μια διεθνή συμφωνία η οποία να είναι, συμ, ε, να είναι δεσμευτική. Εδώ μας λέτε διάφορα καινοτομία, ανανεώσιμες αυτές. Τι θα γίνει όμως όσον αφορά τη συλλογική, την συνολική ε, συμφωνία. Αυτά. Και εγώ μοιράζομαι μαζί σας την ίδια αγωνία. Καταλαβαίνω την ε, αγωνία όσον αφορά τι διαπραγματεύσει για το κλίμα και αυτό που λέτε ότι κάθε φορά ξεκινούμε με ε, πολλές προσδοκίες. Ε, είδαμε το πρωτόκολλο του Κιώτο, είδαμε τη διάσκεψη τη Βαρσοβίας. Έχουμε πολλές προσδοκίες οι οποίες ενθαρρύνονται ε, από την σκέψη ότι μετά από όσα έχουμε δει να συμβαίνουν λόγω της κλιματικής αλλαγής στον πλανήτη, ότι επιτέλους ε, οι κυβερνώντες ε, θα θα πάρουν αποφάσεις. Ε, ε, αυτή τη στιγμή η αύξηση της ε, θερμοκρασίας είναι 0,8. Αν φτάσει αυτή η αύξηση στους δύο βαθμούς τότε οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές. Αλλά ταυτοχρόνως βλέπουμε και άλλα στοιχεία τα οποία διαφοροποιούνται. Ποτέ δεν είχαμε δει τόσες πολλές φυσικές καταστροφές. Ποτέ δεν είχαμε δει τόσο μεγάλες αλλαγές σε πολλές χώρες γιατί έχουν αλλάξει ε, λόγω της γενικότερης ε, αλλαγής, ε, κλιματικής αλλαγής πολλά πράγματα και στην Ασία και στην Ευρώπη. Πιστεύω λοιπόν ότι τώρα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου έχουμε πλέον αυτή την κριτική μάζα στοιχείων και τεκμηριώσεων ότι δηλαδή η κλιματική αλλαγή μπορεί να οδηγήσει σε πολύ αρνητικά στοιχεία, ότι μπορεί να έχει πολύ υψηλό κοινωνικό και οικονομικό κόστος και έχουμε όμως ε, και τα μέτρα και τις δυνατότητες τις τεχνικές έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε ε, την κλιματική αλλαγή. Πιστεύω λοιπόν ο, επίσης ότι ε, βλέπουμε και κάποιες θετικές εξελίξεις σε χώρες όπως οι Ηνωμένες και η Βραζιλία. Γι' αυτό πιστεύω ότι εάν ακολουθήσουμε μια σωστή τακτική αυτή τη φορά θα μπορέσουμε να επιτύχουμε ένα φιλόδοξο συνολικό δεσμευτικό ε, ε, πρόγραμμα. Ο κύριος Κόφοντ. Σας ευχαριστώ πολύ. Εδώ είμαι. Κύριε υποψήφια αντιπρόεδρε, νομίζω ότι μας έχετε δώσει πολύ καλές απαντήσεις απόψε για το πώς να προχωρήσουμε σε μια πράσινη ενεργειακή ένωση στην Ευρώπη. Αλλά είπατε ότι πρέπει να είμαστε οι πρώτοι σε επίπεδο ανανεώσιμων ενεργειών στον κόσμο ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δείτε τις παγκόσμιες επενδύσεις για την καθαρή ενέργεια έχουν μειωθεί σε παγκόσμιο επίπεδο στη Γερμανία, στην Ιταλία και σε άλλες χώρες έχουν μειωθεί σημαντικά αυτές οι επενδύσεις. Πρέπει να ξέρω λοιπόν τι <clears throat> πιστεύετε και πώς θα δράσετε συγκεκριμένα ώστε η Ευρώπη να γίνει το νούμερο ένα σε παγκόσμιο επίπεδο για ανανεώσιμες ενέργειες. Τι σημαίνει αυτό, ποιοι είναι οι δομικοί λύθοι αυτής της πρωτοπορίας, πώς μπορούμε να συγκριθούμε με τον υπόλοιπο κόσμο, πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό, ποιος είναι ο στόχος μέχρι το 2030 όταν τον συγκρίνεται με την πραγματικότητα. 27% για ανανεώσιμες ενέργειες είναι φιλόδοξο στόχος για εσάς. Θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η δική σας θέση. Ευχαριστώ πολύ για το ερώτημά σας. Νομίζω ότι η Ευρώπη είναι ηγέτη σε παγκόσμιο επίπεδο για τις ανανεώσιμες ενέργειες. Γιατί αν δείτε το γεγονός ότι 41% των νέων εγκαταστάσεων για ανανεώσιμη ενέργεια στον κόσμο <clears throat> λαμβάνουν χώρα στην Ευρώπη, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν δείτε την ποιότητα της τεχνολογίας μας Κανείς δεν διαφυσβητεί ότι είμαστε οι πρώτοι στον κόσμο. Και αν δούμε τώρα και την επιχειρηματική πλευρά της ποιότητας αυτής, της τεχνολογίας μας, της πράσινες τεχνολογίες, όλα αυτά καταδεικνύονται από, τον, ε, από την απασχόληση που δίνει ο τομέας αυτός, την ικανότητα να εξάγουμε σε παγκόσμιο επίπεδο, το ότι είμαστε ανταγωνιστικοί και μπορούμε να εξάγουμε αυτές τις πράσινες τεχνολογίες. Πιστεύω λοιπόν ότι τα επόμενα πέντε χρόνια θα δούμε να φτάνουμε σε μία, αν θέλετε, κρίσιμη μετάβαση. Θα πετύχουμε την κρίσιμη αυτή μάζα και θα μπορέσει να μειωθεί το κόστος παραγωγής για τις ανανεώσιμες ενέργειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα μειωθεί λοιπόν σημαντικά. Αν συνεχίσουμε λοιπόν και βελτιώσουμε ακόμα περισσότερε τις τεχνολογίες, αν δούμε πώς μπορούμε να συνδέουμε τις ανανεώσιμες ενέργειες στο δίκτυό μας και αν ξεπεράσουμε τα σημεία συμφόρησης, μπορούμε έτσι να υποφελθούμε πολύ περισσότερο από την ενέργεια, τις ανανεώσιμες ενέργειες, όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε διεθνές επίπεδο και αυτό είναι το βασικό επιχείρημα που εξηγεί ότι πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι για την ανανεώσιμη ενέργεια και αυτό θα οδηγήσει στην επίτευξη ενός στόχου 27% και περισσότερο από 27% γιατί η εμπειρία μας με τις επιχειρήσεις και την τεχνολογία θα μας οδηγήσουν σε πολύ περισσότερη χρήση ανανεώσιμων από 27% κύριος Βέρνετ Λάγκελ. Κύριε Σέρκοβιτ. Δεν απαντήσατε ουσιαστικά το ερώτημα τη κυρία Κιώστιγκερ για το ποια θέση πήρατε όταν αποφάσισε ο κύριος, όταν πρώτο ο Αλμούνια να πάρουμε, πάρει η Επιτροπή μια θέση για το χίκλεπον. Ψηφίσατε υπέρ ή κατά. Δεν πρόκειται για τη θέση σας για την πυρηνική ενέργεια. Μιλάμε για μια τεράστια στρέβλωση ανταγωνισμού. Πάνω από 35 δισεκατομμύρια χάνονται για την Ευρώπη γιατί υπάρχουν εγγυήσει για τιμή πυρηνικής ενέργειας πολύ πάνω από τις τιμές αγοράς. Μιλάει τώρα η Κομισιόν για βιοκαύσιμα προ τη γενιάς που θα υποστηρίζεται μέχρι το 2020. Έχετε και την οικολογική σχεδίαση. Αλλά τι κάνετε με την Γαλλία, τι θα κάνετε με τη Γαλλία, μαζί ζητήσει τα ίδια πράγματα όπως η Μεγάλη Βρετανία για την πυρηνική ενέργεια. Ουσιαστικά λοιπόν φεύγει από το παράθυρο όλη η στρατηγική σα για την ανανεώσιμη ενέργεια, αν συμβεί κάτι τέτοιο. Πώς θα εξασφαλίσετε λοιπόν μια συνεκτική ενεργειακή πολιτική στην Ευρώπη όταν ήδη σε μια τέτοια περίπτωση όπως τη Μεγάλη Βρετανία έγινε ένα τόσο μεγάλο σφάλμα. Αυτό έγινε μετά από την εκλογή του Γιούγκερ και όχι πριν κιόλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την στεναρή αυτή δήλωση που κάνετε. Αν ξανάφουμε και πάλι σε μια περίπτωση όπως το, η περίπτωση του Χίνκλεϊ. Σας λέω ότι αυτό δεν ήταν ένα θέμα που αντιμετωπίστηκε ως θέμα ενεργειακών επιλογών. Ήταν ένα θέμα ανταγωνισμού και αντιμετωπίστηκε από τους κέριους οικονομολόγους της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού και ήταν σαφές εδώ ότι μιλούσαμε για τον κίνδυνο μιας αστοχία στην αγορά και ότι ήταν απαραίτητη η κρατική βοήθεια για να διατηρηθεί. Ναι, και αν με ρωτάτε, εγώ ψήφισα υπέρ αυτού του μέτρου, γιατί θεώρησα ότι ήταν πλήρε συμβατό με του κανόνε ανταγωνισμού για τι κρατικέ επιδοτήσει και σε αυτή την περίπτωση εάν δεν σεβόμασταν τους κανόνες ανταγωνισμού που προέρχονται από τις συνθήκες, η Κομισιόν δεν θα δεχόταν, δεν θα εφάρμοσε σωστά τη συνθήκη και όλα αυτά που προδιαγράφει για τις κρατικές επιδοτήσεις. Για τα βιοκαύσιμα, ο λόγος για τον οποίο εμείς δεν θέλουμε να συνεχίσουμε με τους στόχους για τα βιοκαύσιμα ως το 2020 είναι γιατί απογοητευθήκαμε την πρώτη γενιά βιοκαυσίμων που είχαν ε, συνέπειες απρόβλεπτες. Με τον τρόπο αυτό ουσιαστικά ε, ουσιαστικά εκτόπισαν την παραγωγή τροφίμων για να γίνει παραγωγή βιοκαυσίμων. και τα καύσιμα αυτά και η παραγωγή τους της πρώτη γενιάς δεν είχαν τα αποτελέσματα που προσδοκούσαμε σε επίπεδο μείωσης των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακος. Επομένως, οι προτάσει μας για την έμεση αλλαγή χρήσης γης, το iLook, και να μπορούμε να έχουμε καλά αποτελέσματα σε αυτό το θέμα ε, είναι προτάσει που θα πρέπει να υποστηριχθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη υποστήριξη στη δεύτερη γενιά βιοκαυσίμων. Ναι, ε, κύριε Σεύκοβιτς, Βρισκόμαστε σε μια μεταβατική περίοδο από το παλαιό σύστημα ενέργειας με τα μεγάλα ε, εργοστάσια παραγωγής ενέργειας, ε, πυρηνικής ενέργειας, τα, στις ανανεώσιμες ε, πηγές ενέργειας. Ε, βεβαίως εδώ υπάρχουν πολλές τριβές σε ορισμένε χώρες. αυτοί που χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα επιθυμούν επιδοτήσεις για τη λειτουργία των εργοστασίων τους πώς, ε, θα, πώς μπορείτε να εμποδίσετε ότι υπάρχουν 28 τέτοια εργοστάσια που ζητούν επιδοτήσεις. Δεύτερον, όσον αφορά την ενεργειακή αποδοτικότητα, χαίρομαι που υπερασπιστήκατε την ε, οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό, γιατί εδώ υπάρχει ευρύ πεδίο για ε, λαϊκισμό και δημαγωγία. Ε, η πρόταση, ε, η Επιτροπή έχει προτείνει και 17 άλλα προϊόντα για να συμπεριληφθούν ε, στην ρύθμιση του, του eco-design. Σας ευχαρι... συμφωνείτε με αυτές τις προτάσεις. Απάντηση. Πράγματι βρισκόμαστε σε μια μεταβατική φάση και στρεφόμαστε προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Υπάρχουν χώρες ε, που έχουν ε, πολύ ηλιοφάνεια και αιωλική ενέργεια. Ε, από την άλλη η συσσόρευση ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί, η συμφόρηση της ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα όπως τη Γερμανία, την Πολωνία και τη Σλοβακία, προβλήματα στο δίκτυο δηλαδή. Ε, θα πρέπει να υπάρξει καλύτερη συνεργασία όσον αφορά τη διαχείριση των συστημάτων ε, μετάδοσης ε, ενέργειας, ούτως ώστε να μην υπάρχουν αυτές οι διακυμάνσεις στο ενεργειακό δίκτυο. Γιατί, και πιστεύω ότι αυτό είναι επίσης ένα στοιχείο κλειδί για μια καλύτερη ολοκλήρωση και συμπερίληψη ανώσιμων πηγών ενέργειας στο σύστημά μας. ε, ε ε, θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια εξορρόπηση στα δίκτυα όσον αφορά το eco-design και τη σχετική οδηγία νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να συνεχίσουμε αλλά με έναν έξυπνο τρόπο δηλαδή να βασίσουμε τις προτάσεις μας σε πολύ στέρεες ε, επιστημονικές αναλύσεις και να εμπιστευτούμε μόνο και τους τομείς όπου είμαστε σίγουροι ότι τα αποτελέσματα θα είναι θετικά, θα υπάρχει προσθέμενη αξία και θα αξίζει τον κόπο να το κάνουμε. Ε, και ε, επίσης το εξή. Αυτό που χρειαζόμαστε εδώ είναι πιο έντονες ε, διαβουλεύσει με τους πολίτες. Ακριβώς λόγω του όγκου γραφειοκρατίας και λόγω του στόχου εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης του κόστους για τους πολίτες. Ο κύριος Νούνο Μέλου, τελευταία ερώτηση. Κύριε Υποψήφιε Επίτροπε, υπάρχουν πολλές απειλές για την ενεργειακή ασφάλεια σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει η τροφοδοσία με φυσικό αέριο, τρομοκρατικές επιθέσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θεωρεί ότι πρέπει να καλύπτει μονάχα λιγότερο από το 50%. Ένα μεγάλο μέρος από τις ενεργειακές ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, καλύπτονται από εισαγωγές και φτάνει η συνολική, το συνολικό κόστος σε περίπου ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Ποιοι είναι οι μηχανισμοί λοιπόν σε ένα τρισεκατομμύριο ασφάλειας που προβλέπεται για την ε, δια, διαμετακόμιση φυσικού αερίου. Όταν ξέρουμε τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στην Ιβρική Χερσόνησο, θεωρείτε ότι είναι δικαιολογημένε οι επενδύσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν ή όχι. Thank uh, Σας ευχαριστώ. η ε, ενεργειακή αποδοτικότητα. Ε, είδαμε ε, ε, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τεστ αντοχής ότι είμαστε σε καλύτερη θέση, σε πιο ισχυρή θέση από ό,τι πριν από πέντε χρόνια. Ωστόσο και πρέπει και, μπορούμε αλλά και πρέπει να βελτιώσουμε την κατάσταση. Θα πρέπει να δούμε βεβαίως και ποια είναι τα εθνικά προγράμματα, ποια είναι, αν υπάρχει υπάρχει συμβατότητα μεταξύ των εθνικών προγραμμάτων. Επίσης να δούμε τι δυνατότητες αποθήκευσης ε, ε, ε, έχουμε γιατί και εδώ μπορεί να υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης και εν πάση περιπτώσει τα ε, κυρίαρχα ε, ζητήματα και τα κυρίαρχα στοιχεία όσον αφορά τις διαμεθοριακές συνδέσεις, όσον αφορά τις ανάδρομες ροές. Όλα αυτά θα πρέπει να ληφθούν ε, υπόψη έτσι ώστε να βρούμε και να δημιουργήσουμε ένα διασυνδεδεμένο δίκτυο που θα είναι σε θέση να βοηθήσει όποια χώρα αντιμετωπίζει προβλήματα. Τα επίγοντα σχέδια τα οποία, στα οποία αναφέρεστε είναι σχέδια τα οποία έχουν ε, ήδη καταρτιστεί και από τις ε, χώρες ε, μέλη. Όσον αφορά τώρα τα προγράμματα κοινού ενδιαφέροντος για τις περιοχές αυτές οι οποίες συμπιέζονται, οι οποίες πιέζονται περισσότερο ε, νομίζω ότι αρχικά η διευκόλυνση Connecting Europe όντως ήταν πολύ πιο ε, φιλόδοξη και είχε και μεγαλύτερη προβλεπόμενη χρηματοδότηση. Εν πάση περιπτώσει τώρα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες ε, και να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε και την βοήθεια των ε, ε, ιδιωτικών ε, φορέων έτσι ώστε και στην, στις διασυνδέσεις του ηλεκτρικού και του φυσικού αερίου να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Πολύ ωραία. Μετά από την τελευταία απάντηση θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες στη σημερινή συζήτηση για τις ερωτήσεις τους. Να ευχαριστήσω βεβαίως ε, και τον υποψήφιο επίτροπο και αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα τώρα να ε, δώσω το λόγο στον υποψήφιο ε, αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτσι ώστε να κάνει την τελική του τοποθέτηση η οποία δεν θα πρέπει να υπερβεί τα πέντε λεπτά.